κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ξεκινά. Λίγη. με μεγάλη πλειοψηφία 42 υπέρ, 5 κατά, 3 αποχές. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε και την προφορική ερώτηση επίσης ηλεκτρονικά. Έχουμε επίσης ηλεκτρονική ψηφοφορία για την, για την προφορική ερώτηση. Λίγη. 26, 46 ε, ναι, καμία αρνητική ψήφος, δύο αποχές. Ε, συγχαίρουμε ε, την κυρία Γκροστέτ και όλες αυτές οι οποίες συνέμπραξαν. Και τώρα απευθύνομαι στη γραμματεία για την προετοιμασία και θέλω να την ευχαριστήσω και ερχόμαστε στο επόμενο ο θέμα της ημερησίας διάταξης που είναι πώς θα αποφευθεί η σπατάλη τροφίμων, η συγγήτρια Ιάννα Ρόσμπαχ. Έχετε επίσης τον κατάλογο ψηφοφορίας που ξεκινά με την πρώτη συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρώτη και η δεύτερη τροπολογία ε, θα ψηφιστούν μαζί γιατί είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 και 5 είναι συμβατές υπέρ κατά με συγχωρείτε δεν είναι συμβατές πρώτο ή 4 ξαναξεκινάμε λοιπόν ποιος είναι υπέρ της τέσσερα. κατά αποχές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 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά 13 ε, και 14 ε, υπέρ κατά αποχές επίσης καταπίπτουν 14 δεύτερο μέτρο, ε, μέρος. Ποιος είναι υπέρ. Διότι εδώ υπάρχει χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος της 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ Κρατά αποχές εγκρίνεται 18 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές <coughs> επίσης εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά ηλεκτρός, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 36 λίγη εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πενήντα εννέα δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 62 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 63. Λίγη. Απερίφθη. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος λίγη Ναι, τσίμα τσίμα, αλλά υπερψηφίστηκε. 89. Πρώτο μέρος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίνεται και ερχόμαστε τώρα στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. 38 υπέρ, κανείς κατά, 15 αποχές και ε, συγχαίρουμε την Άννα Ρόσμπαχ για την έκθεση αυτή για την ε, αποφυγή των ε, απορριμμάτων στην διατροφική αλυσίδα. Και τώρα ερχόμαστε στο σημείο 10 της ημερησίας διατάξεως, ενεργειακή απόδοση και η νέα οδηγία με εισηγητή τον Πίτερ Λίζε στον οποίο ε, δίδω τον λόγο για να παρουσιάσει μια πολύ σημαντική έκθεση για την κλιματολογική προστασία και για την αποδοτικότητα των πόρων. Όποιος δεν θέλει να παρακολουθήσει αυτή την έκθεση παρακαλώ να εξέλθει αθόρυβα από την αίθουσα και θα περιμένουμε ακόμη ένα λίγα δευτερόλεπτα μέχρι ότου αποχωρήσουν όσοι δεν θα παραμείνουν. So. Λοιπόν, νομίζω ότι ηρέμησε η κατάσταση και δίνω τον λόγο στον Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους θα ευχαριστήσω τους συναδέλφους επίσης ε, εάν σιωπήσουν. Και καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για τις πολλές τροπολογίες, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και για την Επιτροπή ε, Περιβάλλοντες και είναι εξαιρετικές ιδέες τις οποίες μπορούμε να προωθήσουμε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα βασικό ε, στοιχείο τα οποία ήδη συζητήσαμε ε, χθες και η Επιτροπή ξεκινά με, το σκεπτικό ότι ο στόχος της ε, εξοικονόμησης 20% ενεργείας θα μπορέσει να επιτευχθεί όπως είχε αποφασιστεί το 2007. Υπάρχει μία σειρά τροπολογιών ε, είτε για να εντείνουμε είτε να αποδυναμώσουμε το στόχο αυτό αλλά πιστεύω ότι θέλουμε να βοηθήσουμε και τον Chris Davis και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε το στόχο που κατήρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007. Πρέπει απλούστατα να βελτιωθεί για να υπάρξει πλήρη εξοικονόμηση σε σχέση με το 2007. Σε αυτό που βλέπουμε εμείς, διότι η Επιτροπή είχε προβλέψει ε, ένα στόχο βάση προβλέψεων με 68 εκατομμύρια τόνους άνθρακα τους οποίους θα εξοικονομούσαμε οπότε ε, ουσιαστικά σε απόλυτους αριθμούς θα έπρεπε η μείωση να είναι 12,9% ενώ μιλάμε ε, για ένα πιο ρεαλιστικό στόχο τον οποίο θέλουμε να διαγράψουμε για τα κράτη-μέλη και γι' αυτό δεν θέλουμε να είμαστε υπερβολικά αυστηροί αλλά θα θέλαμε έναν σχετικό στόχο, ένα στόχο ενεργειακής ε, παραγωγικότητος διότι αυτό πλέον ε, θα οδηγούσε σε μια καλύτερη κινητοποίηση των ε, τοπικών κοινωνιών. Γι' αυτό και θα μείνουμε στους αριθμούς του συμπεφωνημένους. Επίσης όμως πολλοί συνάδελφοι μας είπαν ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με το carbon leakage και βρίσκω ότι η πρόταση ορισμένων συναδέλφων είναι πολύ καλή σχετικά με την τροπολογία 33 και 34 του Σόνι Γκαρντίνη και άλλων που λέγουν ότι πρέπει εδώ να προσέξουμε ιδιαιτέρως τις, τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν εντατικά ενέργεια και να μην τοποθετήσουμε ένα το όριο ε, και να αφήσουμε το θέμα αυτό στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Επίσης από τις τροπολογίες διαπιστώνω ότι εν μέρη υπάρχει μία πιο αυστηρή αντιμετώπιση της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αλλού μεγαλύτερη ευελιξία. Ε, ιδίως το άρθρο 1, 3, 19 όπου καταρτίζονται οι εθνικοί στόχοι και ε, υπάρχουν και διευκρινήσεις τις οποίες εγώ τουλάχιστον στηρίζω διότι αυτό που θέλουμε είναι στο τέλος να επιτευχθεί ο στόχος μας. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο άρθρο 4, στόχος 3% για τα δημόσια κτίρια. Ε, τέλος πάντων σε διάφορα άρθρα υπάρχουν διάφορες τροπολογίες που ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε, να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι που μπορούν μπορούν να επιτευχθούν και πού μπορεί να επέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν τα κράτη-μέλη δεν είναι στο σωστό δρόμο ε, συνδυάζοντας με μεγαλύτερη ευελιξία στα μέτρα. Ο συνάδελφος Ζίμπερ έχει προτείνει αυτή την οδό και ζητά έναν δεσμευτικό στόχο για τα κράτη-μέλη κατά τρόπον ώστε να επιτύχουμε τα 20% σε σχέση με τις προβλέψεις και ε, ένα άρθρο προτείνει να το διαγράψουμε τελείως. Μπορώ να αντιληφθώ ότι αυτό ίσως να είναι μια καλή λύση και το συζήτησα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την προηγούμενη εβδομάδα αλλά αντιλαμβάνουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να ακολουθήσουν αυτή την οδό γι' αυτό και πρέπει να ζητήσουμε να γίνουν πιο αυστηροί εθνικοί στόχοι και να υπάρξει ευελιξία των κοινοτικών ε, μέτρων που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα το κοιτάξουμε και ήδη σήμερα το απόγευμα θα έχουμε την πρώτη συζήτηση. Ε, σε θέματα που είμαστε αποκλειστικά αρμόδιοι, τι θα γίνει με, το effort sharing, την, ε, τον καταμερισμό της ε, προσπαθίας, θα αφαιρεθούν προϊόντα από την αγορά και θα υπάρξει ε, μία επέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να σταθεροποιηθεί το κόστος του πιστοποιητικού και χθε συζητήσαμε με τον Chris Ντέιβις τα θέματα αυτά. Εγώ δεν συμφωνώ με μία τόσο ριζοσπαστική πρόταση και πιστεύω ότι θα έπρεπε να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο και προτείνω να ζητήσουμε κάτι ε, πιο συγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να παρακολουθήσει αυστηρά την αγορά, διότι αν αυξήσουμε το κόστος του πιστοποιητικού και έχουμε ύφεση θα υπάρξει μείωση και να επιτύχουμε μια ενεργειακή αποτελεσματικότητα κατά τρόπον ώστε οι επιχειρήσεις οι οποίες απειλούνται να μην επιβαρυνθούν. Θα πρέπει λοιπόν να αναθέσουμε σαφώς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ένα συγκεκριμένο στόχο χωρίς να την επιβαρύνουμε. Ε, Συζήτησα και με έναν ειδικό και θεωρώ ότι πολλά μέτρα δεν αναφέρονται στο ETS αλλά στο effort sharing, στον καταμερισμό της προσπαθίας και ε, θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει ένας νέος καταμερισμός των προσπαθειών. Συζητώ επίσης όλοι να προωθήσουμε την προσπάθεια διευκρινήσεως με την Ήτρε. Έχουμε ζητήσει συνεργασία με την Επιτροπή αυτή και ε, η συνεργασία δεν προχωρά στον τρόπο με τον οποίο θα θέλαμε να ε, προχωρήσουμε και ε, θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα προωθήσουμε τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν διατυπώσει τροπολογίες. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, ε, ιδίω για πολλά θέματα και ε, ίσως ε, θα έπρεπε να προσπαθήσουμε ε, να καταλήξουμε ιδίως εάν υπάρξουν συμβιβαστικές λύσεις οι οποίες προτιμηθούν. Ευχαριστώ τον Πίτερ Λίζε, θα ψηφιστεί τον Ιανουάριο και στην ε, Επιτροπή του Δεκεμβρίου στην Επιτροπή. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ για την εργασία ε, διότι υπάρχουν 440 τροπολογίες και φαντάζομαι θα καταλήξουμε σε πολλές συμβιβαστικές. Τώρα όμως έχουμε ε, τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι θα επέμβουν. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή και πιστεύω ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί ακόμη και αν έχουμε 440 τροπολογίες μπορούμε να καταλάβουμε και ιδίω από τη συνεργασία με τον ο συντονιστή ότι θα καταλήξουμε ε, σε ε, συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες ποιοτικά θα είναι πολύ υψηλέ. Θέλω εδώ να σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητες των ε, σοσιαλιστών, ε, ιδίω η πρόβλεψη, διότι θα πρέπει να συμμετάσχουν όλες οι ομάδες και διαφορετικά δεν θα υπάρξει πρόοδος του συστήματος Δηλαδή υπάρχουν ε, και άλλες προτεραιότητες ε, οι οποίες ε, δεν αναφέρονται εις τη νεολική ανέργεια αλλά στα smart meters πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις εργατικές κατοικίες και το θέμα της ενεργειακής φτώχειας που αναφέρεται σε αυτή την ε, οδηγία. Ευχαριστώ για τις ε, ε, τροπολογίες οι οποίες ζητούν να ενημερωθούν πλήρως οι καταναλωτές διότι εμείς είμαστε αντίθετοι όλη η οδηγία να απορριφθεί. Μια τέτοια πρόταση έχει υποβληθεί σαν τροπολογία και ε, θεωρώ ότι ο συνάδελφος Ζέμπερτ έχει διαγράψει μία σωστή πρόταση για το μέλλον και θα μπορέσει να υπάρξει μία συμβιβαστική τροπολογία με την Επιτροπή επ' αυτού. Ευχαριστώ. Ο Μύρος Λαφούτσκι τώρα. Ευχαριστώ. Έχω να σας πω τα εξής. Η δικιά μας πολιτική ομάδα στηρίζει ολόκληρη αυτή την ε, ε, οδηγία γιατί πιστεύω ότι μόνο έτσι θα επιτύχουμε μία αποτελεσματική Ευρώπη και σας είχα πει πάντοτε ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε την Ευρώπη και δεν πρέπει να την επιβαρύνουμε. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να απορρίψουμε στο σύνολό της την οδηγία αλλά έχουμε ένα πρόβλημα με τους ε, δεσμευτικούς στόχους ακόμη και αν είμαστε μειοψηφία σε αυτή την Επιτροπή διότι θα υπάρξει ε, αντίδραση από το Συμβούλιο και όσον αφορά τους στόχους άκουσα τα σχόλια, διάβασα τους ε, ε, τα σχόλια του Business Europe και πρέπει να πω ότι βλέπω ότι εις την πρόταση του συναδέλφου Λίζε το 3% που αναφέρεται ή στην ανακαίνιση των ε, κτηρίων είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνομαι αλλά θα δεσμεύσει μεν δημόσιους πόρους για τις επιχειρήσεις αλλά δεν ξέρω ε, αν σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία στη σημερινή συγκυρία θα μπορέσουν να σεβαστούν έναν τέτοιο στόχο χωρίς να αυξήσουν ε, το δημόσιο χρέος τους. Οι πάρα πολλές α, ε, τροπολογίες άλλωστε αποδεικνύουν ότι αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική και εγώ είμαι της άποψης ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να προχωρήσει ε, με σωστό τρόπο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ ο Καρλ Στέτερ. Ναι, μιλώ εξ ονόματος του σκιώδη συγητή μας και να ευχαριστήσω τον Πίτερ Λίζη για την πρόταση. Ε, βεβαίως θα καταθέσουμε και εμείς τροπολογίες και οι τροπολογίες σχετίζονται καταρχάς με το συνολικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας, ο οποίος θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι 2% και θέλουμε να αναδιατυπώσουμε και λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει, να μην αποκλείσουμε για παράδειγμα τις μεταφορές. Αλλά το 1,5% θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξο στόχος, ιδίως αν ε, λάβουμε υπόψη και την εξοικονόμηση ενέργειας στον καταναλωτικό τομέα, διότι δεν είναι 100% το ποσοστό εκεί. Εάν ε, ε, εξοικονομούμε μία κιλοβατόρα την ώρα, ε, θα έχουμε μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Επίσης, καταθέσαμε μία τροπολογία που υπολογίζει εκ νέου όλους τους εθνικούς στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, διότι θεωρούμε ότι αυτό το απόλυτο 20% μείωσης είναι ο πραγματικός ε, στόχος που θα πρέπει να επιτύχουμε. Αν έχουμε μία σχετική μείωση σε σύγκριση με ένα βασικό σενάριο, θα υπάρχει πρόβλημα στον υπολογισμό της του βασικού ποσοστού και δεν θα μπορούμε ίσως να επιτύχουμε το στόχο τον οποίο θα έπρεπε να επιτύχουμε για την ε, πολιτική μας, για το κλίμα ο στόχος του απόλυτου 20% είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτύχουμε και άλλους στόχους. Αν καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε λοιπόν χρήματα και εξοικονομήσουμε εδώ θα έχουμε διανύσει πολύ δρόμο. Όσον αφορά τώρα τη σχέση μεταξύ της ε, εξοικονόμησης ενέργειας και του συστήματος εμπορίας εκπομπών, θεωρούμε και έχουμε καταθέσει και μια σχετική τροπολογία μαζί με, σε, με ε, άλλους ο γραμμικός συντελεστής μείωσης θα πρέπει να είναι ε, διαφορετικός γιατί αλλιώς θα έχουμε 1,54 δισεκατομμύρια ευρώ και επομένως ε, θα πρέπει να κάνουμε αυτή την προσαρμογή με το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Αν δούμε τομείς που δεν έχουν εμπορία εκπομπών, ε, θέρμανση και ούτω καθεξής, θα έχουμε πάνω από 40% μείωση των εκπομπών που θα μπορούσαν να προέρχονται από αυτού του τομέου και αυτό φυσικά ε, θα προσθεθεί και στο ποσοστό που θα έχουμε από το σύστημα εμπορία εκπομπών και πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή ε, στην κατανομή των ποσοστώσεων. Να δω αν έχω κάτι άλλο. Α, έχω ήδη εξαντλήσει το χρόνο μου. Καλύτερα που δεν κατάφερα να τα πω όλα, αλλά έχουμε και άλλα, μην ανησυχείτε. Yeah. Δυστυχώς πρέπει να κοιτάξω το χρόνο διότι χθε είχαμε πρόβλημα. Δεν κοιτούσα την ώρα και αντιμετωπίσαμε προβλήματα με το τελευταίο θέμα. Οπότε παρακαλώ όχι πάνω από τρία λεπτά για να μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο. Η Σαμπίνε. Και εγώ καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να του πω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, θεωρεί ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τις θέσεις μας για την πρόθεση των εξύπνων ενεργειών και γι' αυτό σαν πράσινη έχω ε, προσυπογράψει τους ε, στόχους της ενεργειακής εξοικονόμησης και στο άρθρο 6 πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ετήσια δέσμευση μειώσεως κατά 1,5% για την ε, χοντρική και λιανική πώληση και ε, πρέπει να υπάρχει και ένα συνδυασμός με υποχρεωτικά μέτρα που θα ληφθούν από τα κράτη-μέλη και σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ινστιτούτου στη Χάιντελβεργ για την έρευνα της ε, χρήσεως ενεργείας μέχρι το 2014 έτσι θα αποδεσμεύαμε 14 δισεκατομμύρια ετησίως το χρόνο και όσον αφορά τις εισαγωγές ε, ορυκτών καυσίμων θα μπορούσαμε να μειώσουμε το κόστος ε, ανά έτος μέχρι 5,5 δις. Ευχαριστώ, ορέστε. Ο κύριος Ρώση δηλαδή. Θέλετε να μιλήσετε. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, εμείς ε, παρουσιάσαμε αίτηση απόρριψη τη διάταξη αυτή, διότι θεωρούμε ότι είναι πολύ επαχθε και δεν είναι δυνατόν να το προτείνουμε όπως ακριβώς προτείνεται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ε, το άρθρο 6 που αφορά τις υποχρεωτικές ε, ε, πτυχές, ε, διότι επιβαλλούμε ουσιαστικά τα ίδια μέτρα στα κράτη-μέλη. Στο 7 έχουμε τα ίδια στοιχεία, επιβάλλονται τα ίδια συστήματα. Στο 19 έχουμε αντίστοιχα μελλοντικά υποχρεωτικά συστήματα με αναθεώρηση ε, στις 30 Ιουνίου του 2014. Η παράγραφος 5 είναι τροποποίηση ε, άλλων νομοθεσιών που ήδη είναι ενισχύ το EPPC, ακούσαμε και την ομοθεσία για τις μεταφορές ή την πρόταση των πρασίνων να τροποποιήσουμε την κατανομή των ποσοστώσεων στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να αναβάλουμε και θα πρέπει να ξαναγραφτεί από την αρχή, διότι υπάρχουν και κάποια αιτήματα όπως για παράδειγμα εξυγχρονισμός κτηρίων, δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων, οι οποίοι είναι αδύνατον να υλοποιηθούν ιδίω ε, τη δεδομένη στιγμή το να λέμε ότι ε, θέλουμε να έχουμε ένα 3% δημόσια πάρκα και κάποιες ε, άλλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν αδυναμίες εγγενείς να γίνουν σε κάποιες χώρες που έχουν και πάρα πολλούς ιστορικούς χώρους. Ε, η άποψή μας είναι καθόλου επικριτική. Υπάρχουν 1.700 ε, τροπολογίες τρομακτικές από την Αρμόδια Επιτροπή. Ε, κατά την άποψή μου θα έπρεπε να τα ξαναδούμε όλα από την αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτοί ήταν οι σκιώδεις συζητητές και τώρα πάμε στους άλλους ομιλητές, ο Ρίχαρτ Ζέμπερτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Πίτερ Λίζε διότι πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ε, η εξοικονόμηση του πετρελαίου που επιζητείται πρέπει να επιτευχθεί και πιστεύω ότι αυτό είναι το ουσιαστικό θέμα αυτής της προτάσεως ε, και είναι ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο σκοπεύει να το επιτύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς καταρτίζει δεσμευτικούς στόχους αλλά το αποτέλεσμα δεν ακολουθεί τις προσπάθειες πρέπει να πείσουμε τα κράτη να δεχθούν δεσμευτικούς στόχους αλλά να τους πούμε ότι τα μέτρα τα οποία θα τους προταθούν θα είναι ευέλικτα και όπως είπαμε στο άρθρο 8 να υπάρχει αυτή η ευελιξία ε, κατά τρόπον ώστε να επιτύχουμε. Όσο όμως ο πιο δεσμευτικός γίνεται ένας στόχος τόσο περισσότερο είναι το κόστος του και ε, τόσο μακρύτερη θα είναι η διάρκεια του. Οπότε μπορεί να ισχύσει μέχρι το 2013-2014, δηλαδή θα έχουμε χάσει πολύ χρόνο και θα έπρεπε να έχουμε το θάρρος σαν κοινοβουλευτική εδώ να προτείνουμε κάτι διαφορετικό. Διότι τα μέτρα τα οποία προτείνονται ε, δεν με ικανοποιούν. Γιατί αυτά και όχι άλλα. Διότι σε ανατομής έχουμε πολλά. Ε, έχουμε πάρα πολλές ρυθμίσεις και στα κτίρια έχουμε πολλούς στόχους και εδώ μεταφέρουμε και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Είναι κάτι δηλαδή πολύ περίπλοκο το οποίο μας έχει επιβληθεί από την Ευρώπη χωρίς να έχουμε αποτελεσματική χρήση και ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και η πιο απλή λύση θα ήταν να συνδυαστεί με καλή εφαρμογή ε, αντί για ένα πολύ περίπλοκο ε, νομοθέτημα με φοβερή γραφειοκρατική εμπλοκή η οποία δεν θα μας καλύψει. Θα πρέπει οι συνάδελφοι να έχουν το θράρος να μπορέσουν να δεσμεύσουν τα κράτη-μέλη και να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ τον Ρίχαρτ Τζέμπερ. Θα πρέπει ο στόχος ε, να είναι δεσμευτικός αλλά να υπάρχει ευελιξία για το πώς θα επιτευχθεί. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Πίτερ Λίζε όσον αφορά το 3% ε, της ε, διάταξης που αναφέρεται στον περιορισμό ενεργείας των δημοσίων κτηρίων που χρειάζεται αποτελεσματικότητα ενεργείας και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας βλέπουμε ότι ακόμη και εδώ υπάρχουν διαφορετικές ε, καταστάσεις οπότε πρέπει να δούμε τι είναι ένα τέτοιο κτίριο. Υπάρχουν ε, δημοτικά κτίρια όπου υπάρχουν πολλές κοινωνικές κατοικίες που δεν μπορούν ε, να αντιμετωπιστούν αν δεν υπάρχει το αντίστοιχο ενίκιο και αντιλαμβάνουμε ότι παντού υπάρχει ένα πρόβλημα και κατεδαφίζονται πολλά δημογραφικά δηλαδή βλέπουμε ότι δεν συνάδουν ε, τα κτίρια αυτά με τους στόχους του 2030-2040 πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία διότι διαφορετικά οι δημοτικές αυτές επιχειρήσεις θα έχουν πρόβλημα να υλοποιήσουν το στόχο τους. Και τώρα η Φρανσουάς Γκροστέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προτιμούσα να συζητήσουμε για δεσμευτικούς στόχους και όχι δεσμευτικά μέτρα διότι χρειάζονται συμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητος και ε, για να έχουμε καλές συμβάσεις αυτού του είδους θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε σωστούς οικονομικούς ελέγχους. Ελέγχους οι οποίοι πρέπει να γίνονται από εσωτερικούς ε, εμπειρογνώμονες με τα κατάλληλα προσόντα και οι οποίοι φυσικά δεν θα ε, συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες που υπόκειται σε αυτόν τον έλεγχο. Φυσικά υπάρχουν πολύ σημαντικοί τομείς ε, σε αυτό το χώρο της ενεργειακής απόδοσης για την ανακαίνιση ας των κτηρίων και θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι αυτοματισμοί, κάποια ευφυΐα στα δίκτυα ε, διανομής ενέργειας. Πρέπει επίσης να εμπλακεί πολύ περισσότερο ο καταναλωτής. Δηλαδή, Ξέρουμε ότι υπάρχει μια εχμή στην κατανάλωση κάθε βράδυ όταν ο κόσμος επιστρέφει σπίτι του από τη δουλειά και ε, ανάβει κάποιες συσκευές. Πρέπει ο καταναλωτής να συμμετάσχει για να έχει τέτοια συμπεριφορά η οποία θα επιτρέπει πραγματική ε, αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Αυτό που θέτει σε εκείνο τον κλάδο είναι αν δεν μπορούμε να διατηρήσουμε σταθερούς τους κανόνες που ε, θεσπίσαμε όταν ε, θεσπίσαμε το σύστημα ε, των εκπομπών. Γιατί αν αλλάξουν οι κανόνες θα χαθεί η εμπιστοσύνη των παραγόντων και θα δεν θα έχει πια αξιοπιστία το σύστημά μας. Πρέπει λοιπόν ε, να δούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας ε, στην, ε, στον τομέα της σωστής χρήσης της ενέργειας και να μετρήσουμε κάθε δραστηριότητα σε σχέση με την απόδοσή της πρέπει να είναι δυνατόν να προτιθούν, να υλοποιηθούν εναλλακτικά μέτρα που συνεπάγονται παρόμοια προσπάθεια, χωρίς όμως να πρέπει ή να επιτρέπεται ή να αντιτίθεται συστηματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να στοχεύσουμε σε όλους τους επενδυτές, επιβάλλοντας όχι μία τεχνική λύση με συστηματικό τρόπο, αλλά να θεσπιστεί μία αξιολόγηση κόστους αποτελεσματικότητας, όπως επίσης και την κατάλληλη ε, επιλογή του τόπου. Σας ευχαριστώ. Merci ε, Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κυλακάκης. Thank you. There are... Ευχαριστώ. Καταρχάς να πω ότι ο Πίτερ Λίζε έκανε πολλή δουλειά για το ζήτημα αυτό νομίζω καλή δουλειά, αλλά για τρία συγκεκριμένα θέματα, το ένα εξ αυτών είναι η ανακαίνιση δημοσίων κτηρίων. Ξέρουμε ότι έχουμε λιτέτητα, πολύ πιεσμένο προϋπολογισμό και πρέπει να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τα χρήματα των φορολογουμένων. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω, όταν παρεμβαίνουμε, να γίνεται μια ανάλυση κόστους ωφελίας που θα λαμβάνει υπόψη και την μελλοντική αλλά και την τρέχουσα χρήση ενός δημοσίου κτηρίου. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου τα θέματα της ενεργειακής απόδοσης δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με τη χρήση του κτηρίου. Ε, Μπορεί να είναι ένα κτίριο, για παράδειγμα, ένα άδειο κάστρο, στο οποίο θα δαπανίσουμε εκατομμύρια για να είναι αποδετικός προς την ενέργεια και τελικά να μην χρησιμοποιείται από κανέναν. Δεύτερον, όταν γίνεται αγορά ενός νέου κτίριου και λέμε ότι θα πρέπει να είναι ενεργειακά αποδοτικό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλους παράγοντες, διότι η αγορά ενός κτιρίου είναι πολύ σημαντική αγορά για το δημόσιο τομέα Επομένως, θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτή την πτυχή και να μην ε, γίνεται μια αγορά στα τυφλά. Επίσης, οι εταιρείε ενέργειας όταν χρησιμοποιούνται ως προαγωγή ενεργειακής απόδοσης δημιουργούν ψευδή κίνητρα. Οι εταιρείε ενέργειας έχουν κίνητρο να πολλούν ηλεκτρική ενέργεια. Όταν εμείς λοιπόν τους χρησιμοποιούμε για να προωθούμε την ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε ε, τα ψευδή αυτή, ε, τα στρεβλά αυτά κίνητρα να μην αποτελούν και αποτρεπτικό παράγοντα για ανασταλτικό παράγοντα για την ε, αποτελεσματική του εργασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πέτρο Λέζε για την εξαιρετική ανάλυση που έκανε στο θέμα αυτό. Έχω κάποια συγκεκριμένα θέματα που θέλω να θέσω. Είπε ότι πρέπει να σκεφτούμε τα ευέλικτα μέτρα. Είμαι υπέρ. Ξεκινάω από το άρθρο 4, τη δέσμευση για το 3%, του στόχου για τα δημόσια κτίρια. έχει διατυπωθεί ότι θα πρέπει κάθε χρόνο να ανακαινίζονται το 3% των κτηρίων και αυτό επαφείται στις τοπικές αρχές. Μιλάμε δηλαδή για την ε, κοινωνική στέγαση. Θα γίνει μεγάλη αύξηση των ε, ανακαινήσεων. Και γι' αυτό στην τροπολογία μου λέω ότι αντί να αναφέρουμε αυτό το ψηλό ποσοστό 3% να πούμε 2% αλλά θα πρέπει να μην ε, ε, επιμείνουμε τόσο πολύ ώστε στο κάθε χρόνο να γίνεται το 2-3% και στην τροπολογία μου 1-1-1 αυτό ε, προτείνω. Να παίρνουμε τους μέσους όρους τώρα, στο άρθρο 10. Τα ετήσια σχέδια θέρμανσης αναφέρονται οι εθνικές διατάξεις που πρέπει να ισχύουν στο, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο χώρας και τα οποία θα πρέπει να ε, ευθυγραμμιστούν με ε, τα σχέδια του κώδικα. Διερωτώ με σε τι θα ωφεληθεί η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Υπάρχουν αρκετά λεπτομερείς διατάξεις ε, χωροταξίας και πολεοδομίας για τις τοπικές αρχές οι οποίες περιορίζουν την ανεξαρτησία των τοπικών αρχών. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η κατάσταση εδώ. Επίσης το άρθρο 10 η πιο ε, αποτελεσματική χρήση της συνδυασμένης χρήσης ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης. Αν υπάρχει μία μονάδα ε, παραγωγής με φυσικό αέριο, δεν χρειάζεται να γίνει αυτός ο συνδυασμός ε, κατά ανάγκη. Θα ήθελα λοιπόν να το δει ο αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα θέματα. Κυρία Βέσλοντ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ενεργειακή απόδοση είναι κάτι το οποίο μας ε, απογοητεύει όλους. Είναι τόσο προφανές αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και τελικώς ε, δεν γίνεται. Το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται μέτρα σημαίνει ότι οι στόχοι πρέπει να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα παρά το γεγονός ότι διαφωνούν τα κράτη-μέλη. Εάν δεν υπάρξουν μεγαλύτερες πιέσεις δεν γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν. Αυτό είναι σαφές. Επιπλέον, όπως είπε και ο συνάδελφος Γιολάινεν, είναι λίγο αντιφατικό να γίνεται ένας ε, τόσο συγκεκριμένος ε, κανονισμός ε, για τους δημόσιους στόχους και από εκεί και πέρα να μην είναι δεσμευτική. Θα πρέπει να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας και όχι να καθόμαστε να αναλύουμε διεξοδικά την ενεργειακή απόδοση των δημοσίων κτίριων. Δεν διαφωνώ, αλλά θα προτιμούσα ένα πιο ευέλικτο σύστημα το οποίο να έχει δεσμευτικούς στόχους σε εθνικό επίπεδο. Κατόπιν, θα έπρεπε οι φιλοδεξίες μας αυτές να σχετιστούν με ένα 5% μείωση ε, εξοικονόμηση ενέργειας. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος τον οποίο θα έπρεπε να ακολουθήσουμε και θα πρέπει να αντλήσουμε και διδάγματα από τα αποτελέσματα των μακροπρόθεσμων στόχων για να μπορέσουμε να έχουμε και προβλέψεις ε, τις οποίες θα δώσουμε σε όλους τους ε, ενεργειακούς τομείς. Να υπάρχουν στόχοι για το 2015, για το 2030 για να μπορέσουν όλοι να προσανατολιστούν λίγο ε, προς το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και βέβαια η Σουηδία είναι χώρα με υψηλό επίπεδο κτηρίων. Το ερώτημα είναι πώς ε, λαμβάνεται υπόψη αυτά το, αυτό το οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα, ενώ αλλού ίσως να μην έχουν γίνει τόσα πολλά. Είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό. Ε, να ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σε σχέση με αυτές που πρέπει να καταβληθούν. Η Κριστίνα Κροτίνος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εμένα αυτή η οδηγία μου δημιουργεί εκνευρισμό σε μεγάλο βαθμό, διότι θεωρώ ότι εμπίπτει σε όλο αυτό το πλαίσιο του τρόπου με τον οποίο νομοθετεί η Ευρώπη. Στο παρελθόν περιμέναμε να οριμάσει μια ιδέα, γινόταν ένα έλεγχο, γινόντουσαν όλα αργά και για να φτάσουμε σε μια οδηγία έχει γίνει μια αρκετή μελέτη. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ε, όπου έγινε κάτι το 2004, τώρα βρήκανε κάποιες αντιφάσεις και τα αλλάξανε το 2009 και τώρα τα ξαναλάζουμε. Και ουσιαστικά είχαμε λάβει υπόψη ε, κάτι το οποίο είχαμε να το εξετάσουμε στο παρελθόν και τώρα φαίνεται ότι αυτό έχει γίνει κανόνας. Εμένα ο στόχος αυτός δεν μου αρέσει. Και γιατί δεν μου αρέσει. Γιατί τώρα ουσιαστικά θέλουμε να είναι υποχρεωτική η ενεργειακή απόδοση στα κράτη-μέλη. Εγώ Εργάζομαι απευθεία με τους ε, υπεύθυνου του κλάδου. Βλέπω τι γίνεται με την ε, ανοικοδόμηση μιας περιοχής η οποία πλήχθηκε από το σεισμό και προσπαθούμε να έχουμε στο μέγιστο δυνατό ενεργειακή απόδοση στα κτίρια. Αλλά υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που δεν συνυπολογίζονται. Για παράδειγμα, στο άρθρο 7 το σύστημα που έχουμε ε, για τα ευφυή e, συστήματα μέτρησης είναι τόσο ακριβά αυτά τα συστήματα που κανένας δεν θα τα αγοράσει. Ποιος θα φτιάξει τα δίκτυα. Πρέπει να είναι ολόκληροι δρόμοι, ολόκληρες γειτονιές. Εμείς στη Λόρκα ε, σχεδιάζουμε γειτονιές όπου κάθε γειτονιά θα έχει μόνο μία μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε από τον πληθυσμό να αναλάβει ηλεκτρική παραγωγή και όχι μόνο να εξοικονομεί ενέργεια, αλλά να παράγει και ενέργεια. Και το θέμα είναι τι θα γίνει από κοινωνική ε, πλευρά. Δεν μπορούμε να κάνουμε επενδύσει σε μία περιοχή και να μην επωφελείται μία ολόκληρη γειτονιά. Ακόμα και το θέμα λοιπόν της νομοθεσίας, της βασικής νομοθεσίας που βασίζεται στην ε, ιδιοκτησία του καθενός και ο καθένας είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού μου, ας βλέπουμε τώρα ξαφνικά ότι πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά και να υπάρχει κοινωνική ισότητα μέσω της ενέργειας όλοι οι γείτονε θα πρέπει να απολαμβάνουν των ίδιων ωφελών. Αλλά αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να υλοποιηθεί, διότι θα πλήξουμε ένα από τα βασικά στοιχεία, τι βασικέ αρχέ, ότι ο καθένα θεωρεί ότι είναι ιδιοκτήτη του σπιτιού του. Εάν πρέπει κάποιο να πληρώσει τον μετρητή τη ενέργεια, που έρχεται από την τάδε χώρα που γνωρίζουν όλοι, που έχει και ένα καλό λόμπι και προωθεί το προϊόν. Εδώ δημιουργείται ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και γι' αυτό ακριβώ μου δημιουργεί και εκνευρισμό. Το θέμα μου φαίνεται υψής της σημασίας, αλλά τα ιστορικά κτίρια, για παράδειγμα, ιστορικά μνημεία. Εγώ είχα καταθέσει τροπολογία για να αποκλειστούν τα κτίρια αυτά. Τώρα έχω καταθέσει τροπολογία για να αποκλειστούν τα κτίρια αυτά. Αλλά αν για κάποιο λόγο δεν περάσει η τροπολογία μου, δεν συμφωνώ ε, και με, ακριβώς με αυτά τα οποία αναφέρονται σε άλλη τροπολογία. Εγώ ζητώ ειδικά μέτρα για να προσθέξουμε τα κτίρια ιστορικής σημασίας. Και συγγνώμη που μακρηγορώ τώρα. Η οδηγία αυτή μας υποχρεώνει να ε, βάλουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν ελέγχους και οι πόλεις που δεν το κάνουν και δεν κάνουν σημαντικούς ελέγχους θα τιμωρηθούν και δεν θα λάβουν ε, ενισχύσεις. Δηλαδή υπάρχουν ιστορικές πόλεις που έχουν σημαντικά προβλήματα και αυτές θα μείνουν ε, χωρίς πρημοδότηση και θα απομονωθούν από το σύστημα. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και να τους περιλάβουμε όλους. Γίνονται έρευνες στην Ευρώπη για τα ιστορικά κτίρια και για τις ε, καλές ε, δυνατότητες που έχουν για μόνωση, γιατί έχουν για παράδειγμα ε, τυχοποιία όταν κατασκευάζονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια με την αρχιτεκτονική δομή. Υπάρχει ε, αρχιτεκτονική, η οποία έχει έτοιμες τους συλλέκτες και τα πάνελ για τη συλλογή ηλιακής ενέργειας. Νομίζω λοιπόν ότι γίνεται έρευνα για την ενεργειακή απόδοση την οποία δεν παρουσιάζεται. Θα ολοκληρώσω. Τα αποτελέσματα είναι ότι σε ιστορικές πόλεις η απόδοση αφενός είναι η τυπολογία της αρχιτεκτονικής και αφετέρου η χρήση του κτηρίου που γίνεται, οι καλές πρακτικές, αλλά συμπεριλαμβάνομαι και τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς πάμε λοιπόν μόνο στις συσκευές υποχρεώνουμε όλους τους πολίτες να έχουν ένα μετρητή FEE ο οποίος θα είναι πανάκριβος και θα στοιχίζει πάρα πολύ στους πολίτες και τελικώς απλώς θα προωθήσουμε ένα λόμπι. Ευχαριστώ, ήμουν ευγενικό γιατί ξέρω ότι παθιάζεστε με τα θέματα αυτά ε, λόγω και του επαγγελματικού σας βίου ως αρχιτέκτονας. <clears throat> <clears throat> E, λοιπόν, εάν ο στόχος του 20% της ενεργικής απόδοσης τήρηθει, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η έκθεση του κυρίου Λίζε περιλαμβάνει εξαιρετικές προτάσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, δεσμεύσεις και όχι μια απλή κατεύθυνση. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν πολλές τροπολογίες, πράγμα το οποίο δεν βοηθάει. Ας πούμε αυτός ο ενεργειακός έλεγχος κάθε τρία χρόνια ή κάθε πέντε χρόνια. Οι έλεγχοι αυτοί στοιχίζουν. Φερρυπίν ε, στην περίπτωση των νοσοκομείων. Απαιτούν τις επισκευές των οροφών κλπ. κλπ. Και μετά από πέντε χρόνια όταν θα εισαχθούν τα πιστοποιητικά, θα πρέπει να δούμε αν τα μέτρα έχουν τελικά επιτύχει το σκοπό τους. Όσον αφορά το 3% των δημοσίων κτηρίων που θα πρέπει να ανακαινίζονται. Σημαντικό είναι αυτό. Όμως τα δημόσια κτίρια δεν ανήκουν πάντα στις κρατικές αρχές ή στις δημόσιες αρχές. Μπαίνει κανείς στο θέμα του σε ποιον ανήκει το κτίριο. Επίσης πρέπει να προσέξουμε κάπως περισσότερο τα ιστορικά κτίρια. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούν να επιτευχθεί αυτός ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης για αυτά τα κτίρια. Ο κ. Πότσο ανέφερε το θέμα της ενεργειακής ένδυας. Αν το κόστος ή ένα μέρος του κόστους τέλος πάντων το φέρει κάποιος άλλος. Δεν θα πρέπει το κόστος αυτός να το ε, φέρει αποκλειστικά ο οργανισμός παροχής ενέργειας, διότι αυτό θα μετακυληθεί κατά ανάγκη στους ε, πελάτες. Ίσως να υπάρχουν ε, κρατικές βοήθειες, κρατικές ενισχύσεις. Θα ήταν ίσως ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Δεν μπορεί κανείς βεβαίως να έχει κρατική ενίσχυση χωρίς να το παραδέχεται. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν οργανισμοί που θα μπορούν να κρίνουν πότε ισχύει αυτή η περίπτωση. Ο μιλητής η Φλόρενς. Ευχαριστώ και εγώ τον ε, κύριο Λίζε. το δικό μου το πάθος είναι η υποχρεωτική στόχη. Στην προηγούμενη ψηφοφορία ήμουν υπέρ των υποχρεωτικών αυτών στόχων, συνειδητοποιώντας βεβαίως ταυτόχρονα ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς ε, όπως ανάβει κάποιος ένα διακόπτη. Είναι μια μακρά διαδικασία η δεσμευτική στόχη. Στο παρελθόν είχαμε προαιρεκτικούς στόχους ε, και τελικώς τι πήραμε, ε, ψυχία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας και στο τέλος θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λογική λύση όπως αυτή που προτείνει ο συνάδελφος Γλίζε. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και το ενδεχόμενο να καθορίσουμε δεσμευτικούς στόχους. Αυτό ίσως ε, θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε μια πιο λογική λύση με το Συμβούλιο. Η περικοπή κατά 1,5% των, ε, της ε, ενεργειακής, ε, της εξοικονόμησης ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. Θεωρώ ότι είναι λογικό για μονάδες οι οποίες παράγουν ενέργεια μέσω άνθρακα και έχουν δύο, τρεις, τέσσερις, το πολύ πέντε πελάτες. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την εξοικονόμηση αυτή και για φυσικό αέριο να πω και κάτι για τους ελέγχους. Οι έλεγχοι είναι καλό στοιχείο, το βλέπω και στο δικό μου τον ε, κλάδο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε ε, και γιατί ποσοστά συζητάμε. Οι μεγάλοι τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, αλλά μια μικρή επιχείρηση που έχει 30-40 ε, μηχανήματα και ηλεκτρικές γεννήτριες. Δεν ξέρω αν γνωρίζει ένας τέτοιος μικροεπιχειρηματίας ε, τι ενεργειακή επόδοση έχει η επιχείρησή του. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει και έναν υπολογισμό με τόνους αγαθών που ε, παράγονται. Η ενεργειακή απόδοση λοιπόν θα προέρθει μέσω συστού ελέγχου, αλλά χρειάζεται και ένας καλύτερος ορισμό. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, αναφερόμαστε σε συστήματα διαχείρισης ενέργειας και υπάρχουν και φορολογικές επιβαρύνσεις και ελαφρύνσεις αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να ε, χρησιμοποιήσουν την οδό του ελέγχου. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν με τα όσα είπε ο συνάδελφο Λίζε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. το όλο αυτό θέμα στόχο έχει την καταπολέμηση της ε, αύξησης της θερμοκρασίας αλλά και την αντιμετώπιση της ε, κακής κατάστασης του πληθυσμού σε σχέση με την ενέργεια, δηλαδή βελτίωση των συνθήκων ζωής και ε, μείωση της εξάρτησης, της ενεργειακής εξάρτησης των νοικοκυριών. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και θεωρώ ότι η ιδέα του περιορισμού και της θέσπισης προτύπων στον τομέα της αποτελεσματικότητας της ενέργειας ενεργειακής απόδοσης είναι πολύ σημαντικά. Εμείς τώρα ως Επιτροπή Περιβάλλοντος στηριζόμαστε στην πολιτική συνοχής και την περιφερειακή πολιτική στο θέμα αυτό. Δηλαδή, γνωρίζετε στο το πλαίσιο του ΦΕΝΤΕΡ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Οικονομικής Ανάπτυξης, ο κανονισμός για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 προβλέπει ένα μερίδιο 20% των 150 ίσως δις ευρώ ε, και ένα ποσοστό θα πάει στην ενεργειακή απόδοση. Δηλαδή η Ευρώπη θα περιορίσει τα κράτη για να βελτιώσει το θέμα αυτό της ενεργειακής απόδοσης. Θα πρέπει όμως και θετικά να προχωρήσει και να πει πέρα από αυτούς τους περιορισμούς η Ευρώπη συγχρηματοδοτεί και συμμετέχει στη χρηματοδότηση όλων των εργασιών που έχουν σχέση με την ενεργειακή απόδοση. Θέλω λοιπόν εκ μέρους της Επιτροπής Περιβάλλοντος να υποβάλω τροπολογίες σε σχέση με αυτόν τον κανονισμό της ε, περιφερειακής πολιτικής για να ε, κινηθώ στην κατεύθυνση αυτό που είπε η κυρία Μπουτήρες κυρία Ιπνέρ για το, την ιστορική κληρονομιά. Είναι ένα ξεχωριστό στοιχείο. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και πρέπει η Ευρώπη μέσω της περιφερειακής της πολιτικής να συμμετάσχει με τη μορφή της χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταία Στρέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη Γι' αυτό άλλωστε δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει και το γεγονός ότι κατατέθησαν τόσες πολλές τροπολογίες για την έκθεση αυτή. Εγώ Είμαι συντάκτρια της γνωμοδότησης για την Επιτροπή Γυναικών. Δηλαδή βλέπω το όλο θέμα από άλλο πρίσμα, αλλά φυσικά με ενδιαφέρουν και όλα τα θέματα της ε, ε, κοινωνικής στέγασης και θεωρώ ότι η προσέγγιση των κρατών μελών για τα θέματα αυτά ε, και για κτίρια τα οποία ε, χρησιμοποιούνται ως εργατικές κατοικίες, ε, τα οποία θα πρέπει να τα θεωρούμε και αυτά δημόσια αγαθά. Ε, δεν θα πρέπει βέβαια να λησμονούμε ότι υπάρχει και οικονομική επιβάρυνση για τους, για τους καταναλωτές. Παραδείγματος χάρη εργατικές κατοικίες τις οποίες διαμένουν οικογένειες με οικονομικά προβλήματα. Ε, υπάρχουν λοιπόν και κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γι' αυτό και θα πρέπει να δημιουργήσουμε δεσμευτικούς και φιλόδοξους στόχους. Διότι εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Ε, νομίζω ότι είναι προφανής ο στόχος αυτός. Στην Πορτογαλία εδώ και πολλά χρόνια είχε... Ε, εγκριθεί νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των δημοσίων κτηρίων με έξοχα αποτελέσματα. είναι προφανές ότι για κτίρια ιστορικής σημασίας, όπως υπενθύμησαν και αρκετοί συνάδελφοι, ε, ιδίως ε, κτίρια τα οποία βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρούμε τη δέουσα λύση. Διότι ε, στην πλειονότητά τους είναι ε, κτίρια τα οποία είναι ιδιωτική ιδιοκτησία, αλλά ακόμα και αυτά που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, είναι πολύ δύσκολο να πούμε εν μέσω κρίσης ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια για να γίνουν οι κατάλληλες μετατροπές ε, προκειμένου αυτά τα ε, αρχαία ή τα ιστορικά κτίρια ε, να είναι ενεργειακά αποδοτικά. Βέβαια είναι ένα στόχος τον οποίο δεν θα πρέπει να διαγράψουμε και εντελώ. Κατόπιν αναφερθήκαμε και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι προφανές ότι εδώ δεν θα πρέπει να τιμωρήσουμε περαιτέρω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αν δεν κάνω λάθος η οδηγία ε, εξαιρεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επομένως ε, υπάρχει μέρημνα για αυτούς. Ολοκληρώνοντας να πω ότι το να περιορίσουμε το κόστος για τον καταναλωτέ ε, είναι ένας από τους εφικτούς στόχους. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριο Λίζε ορθώς ε, έκανε μία σχέση με την ατζέντα για το κλίμα. Θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή έχει σημαντικά ωφέλη και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν θεωρούμε ότι είναι εμπορική συναλλαγή με οικονομικά ωφέλη. Ίσα ίσα θεωρούμε ότι θα εξοικονομήσουμε 34 δισεκατομμύρια, θα αυξηθεί το ΑΕΠ μέχρι το 2020, θα δημιουργούν θέσεις εργασίας και επομένως υπάρχουν ε, σημαντικά ωφέλη και για την ε, νέα όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία που είναι σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούνται ορθώς τα δημόσια κονδύλια και να συμφωνήσω με την ε, ε, Ευρωβουλευτή που αναφέρθηκε στη χρήση των Ταμείων Συνοχής και επίσης θα πρέπει να υπάρχει και ιδιωτική χρηματοδότηση, δανειοδότηση από τράπεζες παραδείγματι. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον κύριο Λίζα για τη γνωμοδότηση, διότι θεωρούμε ότι προσθέτει θετικά στοιχεία στην έκθεσή μας και ε, θα μας ε, βοηθούσε και η υποστήριξη της ε, Επιτροπής. Είναι ενθαρρυντικό για μας. Σε γενικές γραμμές, αυτό που θέλουμε είναι να φτάσουμε στον τελικό στόχο του 20%, ο οποίος συμφωνήθηκε το 2007. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν είναι σαφές ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει συζήτηση για τα μέτρα ε, τα οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση για τα μέτρα και για τους στόχους. Πέραν αυτού, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς εμένουμε στη θέση μας ότι θα πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση δύο ε, σταδίων για την επίτευξη των στόχων. Το πρώτο στάδιο θα πρέπει να είναι η έγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέτρων τα οποία θα μας οδηγήσουν στο 20%. Αν επιτύχουμε το στάδιο αυτό, τότε περιμένουμε στο πλαίσιο αυτών των μέτρων τα κράτη-μέλη εθελοντικά να καθορίσουν προσωπικούς στόχους οι οποίοι θα προσθέσουν σε αυτό το 20% και δεν θα χρειάζεται από εκεί και πέρα να μπούμε στο φαύλο κύκλο των δεσμευτικών στόχων. Ε, το χρησιμοποίησαμε αυτό το επιχείρημα και το είπε και ο κύριος Ζέμπερ και άλλοι, το αναφέραμε και στην ε, ε, εκστρατεία ενημέρωσης και από τα 27 κράτη-μέλη μόνο ένα κράτος μέλος είναι υπέρ δεσμευτικών στόχων και οι υπόλοιποι ε, είναι αντίθετοι και μάλιστα κάποιοι εξ αυτών στεναρά αντίθετοι στους στόχους. Υπάρχει και αυτό το οποίο αναφέρθηκε, ότι θα υπάρξουν δεσμευτικοί στόχοι και τελικώς ε, δεν θα χρειαστούν δεσμευτικά μέτρα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρούμε ότι είναι σωστή η άγουσα αυτή και ε, δεν ε, θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε το στόχο μας. Ο κύριος Λίζε μας επέστησε και στην ε, ε στροπολογίες 3.33 ε, και 3.34 για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι εντός αυτής της προσέγγισης θα προστατεύσουμε και την εντατική βιομηχανία. Ε, θα το εξετάσουμε και θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά το στοιχείο αυτό. Ως προς τα μέσα τώρα, Υπάρχουν πολλές ιδέες που θα μπορούσαμε να σας παρουσιάσουμε, κάποιες οι οποίες αναφέρθηκαν και στη συζήτηση και προέκυψαν και από την ε, συζήτηση και στις 700 ε, ε, τόσες τροπολογίες που κατατέθησαν και εξετάσαμε. Να σταθώ όμω σε αυτά που μας ανησυχούν και όχι να ε, σας αναφέρω με ποια συμφωνούμε από όσα ακούσαμε στις παρεμβάσεις. Τα λέω με τυχαία σειρά. Ο κύριος ε, Πόκ αναφέρθηκε στην ανάγκη να συμπεριλάβουμε και τον τομέα των μεταφορών. Εδώ έχουμε μια παρέλληλη προσέγγιση και η εφαρμογή του οδικού χάρτη των μεταφορών για το 2050 ε, θα μας βοηθήσει να δούμε και πώς θα πάμε. Δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο όμως να έχουμε και μέτρα τα οποία αλληλοεπικαλύπτονται στη συγκεκριμένη διάταξη για να καλύψουμε και τον τομέα των μεταφορών. Ο κύριος Λάινεν αναφέρθηκε στα θέματα ε, του κόστους ανακαίνησης για τις κοινωνικές κατοικίες ε, και αυτό είναι σημαντικό γιατί αναφερόμαστε σε στρώματα χαμηλού εισοδήματος και επομένως ε, το κόστος θέρμανσης των κατοικιών αυτών, αν εφαρμόσουμε τα μέτρα, θα μειωθεί. αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης, αλλά μέσω πρόθεσμα θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε αυτούς τους στόχους. Ε, δεύτερον, αυτό το ανέφεραν αρκετοί, πρέπει να δούμε πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε τα στοιχεία αυτά. Ε, η κυρία Γκροστέ αναφέρθηκε σε ε, υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες ενέργειας και μείωση των στόχων και συμβάσεις κοινωνικής ε, κοινωνικών κατοικιών που είναι ενεργειακά αποδοτικέ, ε, Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε τους στόχου αυτούς χωρίς να δημιουργήσουμε προβλήματα στου ανθρώπους αυτούς. Επίσης η κυρία Γκροστέτ αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη συμμετοχή των καταναλωτών. Ε, κατανοούμε τις πολλαπλές τροπολογίες οι οποίες κατατέθησαν που ζητούν διάφορα στοιχεία γιατί επέλεγαν να κάνουν αλλαγή για να υπάρξει επιπλέον αξία και να υπάρχει και κίνηση στην αγορά. Μακάρι να προχωρήσει και να ενισχυθεί αυτή η πρόταση. Ο κύριος Κυλακάκης αναφέρθηκε στο 3% και είπε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και ποια ε, κτίρια θα ανακαινήσουμε. Νομίζω ότι η πρότασή μας μας το επιτρέπει να το κάνουμε, διότι τα κράτη-μέλη θα επιλέξουν ποιο θα είναι το 3% που θα υλοποιείται κάθε χρόνο και θα πρέπει να επιλέξουν αυτά τα οποία θα έχουν μεγαλύτερα ωφέλη από την ε, ανακαίνιση. στις τροπολογίες ε, εν γέννη έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες για το άρθρο 6, για το σύστημα που το αποκαλεί ο κύριος Λίλζε υποστήριξη για την ε, εξοικονόμηση ενέργειας. Ε, θα μας άρεσε να αλλάξει ο τίτλος θα θέλαμε να δούμε πού έχουμε εναλλακτικέ λύσεις στην παράγραφο 9 στο άρθρο 6 και πού μπορούμε να ε, έχουμε θετικά στοιχεία. Υπάρχουν όμως κάποιες τροπολογίες οι οποίες ουσιαστικά ε, θα βγάλουν όλα τα βασικά στοιχεία από το άρθρο. Αν δεν κρατήσουμε αυτό το στόχο του 1,5% στο άρθρο δεν θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Και μία τελευταία παρατήρηση. Το άρθρο 8 και τα ευφυείς μετρητές. Ε, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ε, και κάποιες τροπολογίες για το τρίτο πακέτο. Δεν χρειάζεται ευφυείς μετρητές για να έχετε καλύτερη τιμολόγηση. Δεν χρειάζεται να πάμε πιο γρήγορα από το τρίτο πακέτο και αυτά από πλευρά μου. Ευχαριστώ. Θέλει και ο Λίζη να πει κάτι. θα είμαι σύντομος. Καταρχήν, θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά τα οποία ε, είπε ο πρόεδρος και ε, να ε, να πω ότι προβήκαμε σε ε, βελτιώσεις διότι έτσι μπορούσαμε να πετύχουμε ένα πιο συγκεκριμένο στόχο. Η εργασία μας βέβαια προχωράει και δεν θα είναι εύκολο να μπορέσουμε να επιβάλλουμε το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό και οι προσπάθειές μας πρέπει να επικεντρωθούν σε, στο να επιβάλλουμε τις δικές μας απόψεις. Έχουμε συγκεκριμένες απόψεις σχετικά με την κατανομή των βαρών στα κράτη-μέλη. Δηλαδή βλέπουμε όλα τα θέματα στα οποία βασίζεται η πρώτες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολιτικά γίνεται ρεαλιστικό το όλο εγχείρημα. Ε, όσον αφορά την κατανομή των στόχων δεν έχουμε ε, σημαντικές ε, διαφορές. Δεν πρέπει όμως να κάνουμε τον στόχο πιο αυστηρό αλλά να τον κάνουμε δεσμευτικό και μετά να υπάρξει ευελιξία. Όπως είπε ο, ο, ο, κύριος Λάινεν και ο κύριος Χιλακάκης. Ο Θόδωρος πολύ σωστά είπε ότι πρέπει να δούμε πόσο θα διατεθούν οι πόροι γιατί σκέφτεται την κατάσταση της Ελλάδος. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη ε, ευελιξία και γι' αυτό ίσως πρέπει να δείτε το, την τροπολογία 4 αλλά χρειάζεται και άλλη ευελιξία και γι' αυτό είπε ο εάν κατεδαφιστεί ένα δημόσιο κτίριο, δεν υπάρχει λόγος τρία χρόνια πριν να το ανακαινήσουμε. Χρειάζεται λοιπόν ένας πιο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός και να βασιστούμε περισσότερο στην ανανέωση και όχι στην ανακαίνιση γιατί εάν ε, ε, ανανεώνουμε ένα κτίριο το οποίο μετά από πέντε χρόνια θα κατεδαφιστεί δεν υπάρχει κανένας λόγος να δαπανίσουμε ε, χρήματα για την ανακαίνιση και ανανέωση και βελτίωση και εξυγχρονισμό. Γι' αυτό και μιλώ στην τροπολογία 4 ε, για ευελιξία την οποία θα χρειαστούμε για τη χρηματοδότηση. Επίσης όσον αφορά αυτά τα οποία είπε η κυρία Γκροστέτ, ε, Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και ενεργειακή φτώχεια και ε, θα πρέπει να ε, περιλάβουμε τα στοιχεία αυτά. Τέλος, όντως πρέπει να επενδύσουμε, αλλά να αξίζει και τον κόπο, διότι πληρώνουμε 400 δισεκατομμύρια το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ενεργειακές εισαγωγές, δηλαδή σχεδόν όλο το κόστος της γεωργικής πολιτικής της κοινότητος. Εάν λοιπόν ε, τσακωνόμαστε εάν η δαπάνη αυτή είναι σωστή για τη γεωργία πρέπει να σκεφτούμε ε, πάρα πολύ σοβαρά το θέμα της δαπάνης των 400 δις για την ενέργεια και να κοιτάξουμε εάν μπορούμε αυτό το ποσό να το μειώσουμε κατά τρόπον ώστε να μπορούμε θυσίως να το χρηματοδοτούμε. Ευχαριστώ. Όπως ελέγχθη θα ψηφιστεί αυτό στις 20 Δεκεμβρίου. Τώρα, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της ΣΟΤΟΧΑΣ για την εφαρμογή της σύμβασης ΜΑΡΠΟΛ για τις ε, εκπομπές θείου που προβλέπει ότι οι εκπομπές θα είναι 0,5% το 2020 για όλους τους τομείς και δύο, στο 2015 ε, θα είναι 1,15% στις ειδικέ προστατευόμενες περιοχές. Ζητώ όλους όσοι θέλουν να πάρουν το λόγο ε, για το θέμα αυτό να μας πούν τώρα να ζητήσουν τώρα το λόγο για να ξέρουμε πόσο χρόνο θα έχει ο κάθε ομιλητής. Ε, δώστε το λόγο και θα, έχω, θα έχουμε κατανομή του χρόνου. Okay. Thank you very much. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, όσο μόλις είπε ο Πρόεδρος, το βασικό θέμα της πρότασης της, αυτής της Κομισιόν είναι η εφαρμογή της απόφασης του IMO να τεθούν όρι, αυστηρότερα όρια στις εκπομπές θείου από τα πλοία. Τα όρια είναι διαφορετικά όπως και ήδη είναι σε κάθε θαλάσσια περιοχή. Ο IMO, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας, έχει ε, ορίσει περιοχές PF που περιλαμβάνουν τη Βόρεια Θάλασσα, την, Βόρεια, ε, την Βαλτική και το, τη Μάχη και Επισήμως και οι ακτές ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις ε, περιοχές που είναι ελεγχόμενες οι εκπομπές. Το όριο του θείου αυτή τη στιγμή για τα θαλάσσια καύσιμα είναι 1%, θα πάει στο 0,1% από το 2015, από την αρχή του 2015 και στις υπόλοιπες θα είναι 0,5% το όριο θείου στη, το 2020. Θεωρώ ότι αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ε, υγείας στο πενταετία αυτή, διότι το ποσοστό της ε, ατμοσφαιρικής μόλυνσης που προέρχεται από τα πλοία είναι εντυπωσιακά υψηλό. Υπολογίζεται ότι 50.000 άτομα κάθε χρόνο πεθαίνουν προώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης που οφείλεται στα πλοία. Και είναι απολύτως σαφές ότι η ναυτιλία έχει αρχίσει να περιορίζει τις εκπομπές της πολύ αργότερα από τους άλλους κλάδους. Κάποιες εκπομπές που στο παρελθόν υπήρχαν στην ξηρά έχουν μειωθεί κατά 90 ή 80% ανάλογα με το ποια θεωρεί κανείς ότι ήταν η αρχική βάση. Στην Αυστηλία όμως αυτό είναι μια προσπάθεια που μόλις πρόσφατα ξεκίνησε. Αν δεν ληφθούν αυτά τα μέτρα Τότε, τη δεκαετία αυτή, οι εκπομπές θείου από την αυτιλία στις θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης θα ξεπεράσουν όλες τις εκπομπές θείου που προέρχονται από την ξηρά, από όλα τα εργοστάσια, της Μονάδας παραγωγής ενέργειας κλπ. κλπ. Άρα, υπάρχουν πολλά σοβαρά επιχειρήματα υπέρ των μέτρων αυτών που συμφωνήθηκαν στον IMO, στον ε, Διεθνή Οργανισμό ε, Ναυτιλίας. Δεν είναι μόνο η επιλογή του καθαρότερου καυσίμου, αλλά είναι και η επιλογή της χρήσης των λεγόμενων πλυντρίδων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό. Φυσικά, το υγροποιημένο ε, φυσικό αέριο είναι και αυτό μια επιλογή, κυρίως για τα νέα πλοία, αλλά βεβαίως χρειάζεται υποδομή για την ε, τροφοδοσία των πλοίων αυτών σε καύσιμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ε, καθαρίσουν οι εκπομπές ε, του ε, διοξιδίου του θείου, αλλά και των οξυδίων του αζότου και του άνθρακα. Υπάρχει κόστος. Η Κομισιόν όμως έχει υπολογίσει ότι η οικονομική αξία των ε, ωφελών στην υγεία είναι πολύ υψηλότερη από το κόστος των μέτρων αυτών, ανάλογα με τον τρόπο που υπολογίζει κανείς την οικονομική αξία των ωφελών στην υγεία, είναι 2 ή και 25 φορές ε, το, το άλλο κόστος. Είναι η πρόταση αυτή ε, γενικά θετική. Θέλω όμως να την ενισχύσω κάποια σημεία τουλάχιστον της πρότασης θα ήθελα να τα ενισχύσω. Οι τροπολογίες που προτείνω ή είναι οι σημαντικότερες από τις τροπολογίες που προτείνω είναι οι εξή. Πρώτον, η παράταση αυτού του 0,1 του ορίου δηλαδή αυτού, η επέκτασή του στα επιβατικά οχηματαγωγά νωρίτερα από ό,τι το προτείνει η Κομισιόν. Δηλαδή η Κομισιόν το προτείνει, ε, προτείνει να δοθεί μια επιπλέον πενταετία. Εγώ προτείνω το 2015 για τις όλες τις κατηγορίες. Όταν συντάχθηκε η τρέχουσα τροπολογική οδηγία, το όριο για τα επιβατικά αυτά πλοία ήταν το ίδιο με όλα τα υπόλοιπα πλοία. Και προτείνω να διατηρηθεί αυτό, να τηρηθεί η αρχή αυτή. Δεύτερη βασική ε, τροπολογία μου. Αυτό το 0,1% ως όριο να ισχύσει σε, όλες, σε όλα τα ε, ύδατα και εκτός της ΠΕΘ. Δηλαδή, να συμπεριληφθεί όλες οι απαιτήσεις το 0,1 το όριο αυτό που ισχύει για τα πλοία και τα χωρικά ύδατα, σε όλα τα χωρικά ύδατα και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του επόμενου έτους η Κομισιόν θα πρέπει να μελετήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για να θεσπιστούν νέοι τομείς ελέγχου των εκπομπών στις ευρωπαϊκές θάλασσες και να αναφέρει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα συμπεράσματα και να υποβάλει προτάσεις. Το τελευταίο μου σημείο είναι ότι θα πρέπει οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων να γίνουν κάπως πιο ευέλικτοι. Εδώ υπάρχει ένα κόστος και ένα κόστος που κυρίως θα το φέρουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, ο κλάδος που έχει τους μεγαλύτερες ε, διαδρομές. <coughs> Θα πρέπει λοιπόν η μετατροπή αυτή να στοιχήσει λιγότερο με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Και επίσης θα πρέπει να διευκολύνουμε αυτή τη μετατροπή με τη χρήση νέων τεχνολογιών, επιτρέποντας ε, να χαλαρώσουν κάπως για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα οι κανόνες για την ε, για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε ο κλάδος να μπορέσει να ε, ενισχυθεί στην προσπάθεια αυτής της μετατροπής και βεβαίως για να βοηθήσουμε να ξεκινήσει η αγορά αυτής της νέας καθαρότερης τεχνολογίας για τα πλοία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κατάλογος των αγορητών. Έχουμε τους τέσσερις ε, σκιώδης και μετά Ηλεκάκης, Ayuso, Florence, Murkunaite, Tatarella, Manner, Τρεμοπούλος, Κούν and Pirillo. Is anybody missing? Μήπως ξέχασα κανέναν? Αν όχι, κλείνει ο κατάλογος. Τρία λεπτά για τους και ηγητές και οι υπόλοιποι από δύο λεπτά και σας παρακαλώ τηρήστε τα χρονικά προευθέρια, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε καιρούς στη συνεδρίαση. Ο κύριος Φιέρνερ καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε διαπιστώνω ότι όταν ε, ξεπερνάμε το χρόνο σας σηκώνονται τα φρύδια. Οπόμενο, όσο καθυστερούμε τόσο πιο ψηλά φτάνουν τα φρύδια σας. Λοιπόν, είναι καλό το θέμα της αντιμετώπισης αυτό. Περιμέναμε το Διεθνή Λαυτιλιακό Οργανισμό να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Επιτέλους το έκαναν. Είναι θέμα υγείας. Είναι ε, θέμα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στην πηγή του. Θα πρέπει να μειώσουμε το θείο στην πηγή του. Και όλοι έχουν δει πόσο προβληματικό είναι αυτό το καύσιμο. Είναι τόσο ε, πικτό που πρέπει κάποιος να το ε, λιώσει τελείως για να το χρησιμοποιήσει. Βέβαια, ο τρόπος που χρησιμοποίησε το, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας δεν είναι και ο πλέον ε, ευφυής. Για να φτάσουμε από το 2,8 στο, ε, στο 0,1 είναι ποσοστά τα οποία είναι λίγο αδύνατα το 2015 και το 2025 στην Νότια Ευρώπη. Ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι ε, συνέπεια των όσων διαπραγματεύτηκαν τα κράτη-μέλη στον IMO, αλλά ε, η προσέγγιση αυτή μπορεί να είναι καλή για τα κράτη-μέλη όταν σκέφτονται ο καθένα στη χώρα του, αλλά δεν ξέρω αν είναι η πλέον κατάλληλη προσέγγιση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, διότι γνωρίζω ότι τα θέματα υγείας είναι πολύ σοβαρότερα στη Νότια Ευρώπη και μπορεί να ακούγεται περίεργο να λέμε ότι η ζωή ενός Έλληνα είναι λιγότερο σημαντική από τη ζωή ενός Δανού, για παράδειγμα. Δεν θα πρέπει να γίνονται πράγματα τα οποία δεν θα είναι εναρμονισμένα σε οδηγίες. Επίσης θεωρώ ότι αν γίνει με λαθασμένο τρόπο, τότε μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτό που δεν επιθυμούμε, δηλαδή να ξαναγυρίσουμε στα ε, ε, φορτηγά οχήματα και στις δαλίκες. Ε, κατανοώ την πρόταση λοιπόν της κυρίας Χάση, αλλά θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα χωρικά έδωτα και θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να φτάνουμε μέχρι την έκταση που μπορούμε να φτάσουμε για να είναι πιο εναρμονισμένα τα πράγματα. Και ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι το 2015 είναι πολύ ε, κοντά. Μπορεί ίσως και να τα καταφέρουμε, αλλά γι' αυτό και ήθελα και το συζητήσαμε λίγο νωρίτερα να υπάρχει περισσότερος χρόνος για να δούμε τις ερωτήσεις. Συναντήθηκα με Φιλανδούς και Σουηδούς παραγωγούς πλυντρίδων, για παράδειγμα. Και ταυτόχρονα είδα ότι υπάρχουν τέσσερις ε, οι οποίοι παράγουν ήδη και ένας εξ αυτών κάνει πωλήσει μόνο. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα αντιμετωπίσει αυτά στην λεγόμενη εργαλειοθήκη. Θα ήθελα να ξέρω πότε θα μας τα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πότε μπορούν να διευκολύνουν και να ε, υλοποιήσουν αυτή την αλλαγή. Και τέλος, ε, ε, γιατί δεν θέλω να ανέβουν τα φρύδια σας κύριε Πρόεδρε, οι περιοχές ελέγχου θα πρέπει να το συζητήσουμε. Κάναμε μια συζήτηση και για τα σωματίδια στην ομάδα μας και είπατε ότι στα κράτη-μέλη θα δοθούν περισσότερε ευθύνε, διότι εμά μα ε, ενδιαφέρει το θέμα τη διαθέσιμότητα καυσίμων και είπατε ότι λίγο πολύ αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Μπορούν όμω, Είπατε και για τι κρατικέ ενισχύσει. Δεν είμαι βέβαιο κατά πόσον το πρόβλημα των κρατικών ενισχύσεων αυτή τη στιγμή είναι οι κανόνε. Τα χρήματα είναι αυτά που λείπουν. Και αν ξεκινήσουν τα ερωτηματικά για τα χρήματα, ίσω θα πρέπει να σκεφτούμε το πότε και όχι το πώ. Ευχαριστώ που σταματήσετε, γιατί αλλιώ θα έπρεπε μετά να κολλήσω σε λοτέιπ στα φρύδια μου. Η κυρία Κράμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν μιλάτε για ένα μέτρο ποιότητος του αέρα, τότε ε, πρέπει να υπενθυμίσω ότι στις απαρίθμητες ρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια το Κοινοβούλιο έχει διακηρύξει ότι δεν χρειάζεται να επικεντρωθούμε τόσο στις πόλεις όπου δεν είμαστε αποτελεσματικοί. Εδώ έχουμε μία ένα μέτρο το οποίο μπορεί να επιτύχει το στόχο μας, να βελτιώσει ε, την ποιότητα των καυσίμων. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ χρήσιμο το μέτρο αυτό, διότι έχουμε κάνει πολλά για πολλές εγκαταστάσεις στη θάλασσα και αλλού υπάρχουν πράγματα τα οποία υπολείπονται ακόμη ε, και ε, γι' αυτό έχει νόημα. Και υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει μία διεθνή συμφωνία διότι όπως και στους άλλους τομείς καλό θα είναι να υπάρχει μία διεθνή συμφωνία υπάρχει ήδη ένα μέτρο το οποίο είναι νομικά δεσμευτικό και δεν μπορούμε να παρακάμψουμε γι' αυτό και καλό θα ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να το εφαρμόσουμε. Υπάρχουν όμως ορισμένα θέματα τα οποία πρέπει να προωθηθούν δηλαδή πέραν της προτάσεως του IMO πρέπει να προχωρήσουμε πολύ παραπέρα. Δεν είναι αυτό το βασικό, δηλαδή αν θα έχουμε παντού 0,1% ποσοστό θείου στα καύσιμα, το θέμα δεν είναι αν, το θέμα είναι πότε και αν θα λειτουργήσει ε, τεχνικά ε, και όσον αφορά τις περιοχές ΣΕΚΑ όπου υπάρχει ο έλεγχος αυτός του θείου πρέπει να δούμε εάν είναι δυνατόν, εάν έχουμε τα ε, όργανα μετρήσεως, αν είναι αποτελεσματικά, δηλαδή δεν νομίζω ότι το γεγονός να ανακοινώνονται νέες περιοχές ΣΕΚ πρέπει να αφαιθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω να αναφέρω και ένα μέτρο ακόμη, δηλαδή δεν είμαι ευρωβουλευτής ε, δεν έρχομαι από μία εμπλεκόμενη περιοχή ε, και πρέπει να αναρωτηθούμε αν στις περιοχές ΣΕΚ όπου υπάρχουν ε, μεταφορές μικρών αποφάσεων, αποστάσεων, δηλαδή φέριμποτ ή ακτοπλοϊκά. αν οι επιπτώσεις αυτής της νομοθεσίας δεν θα είναι άδικες, δηλαδή αν δω το ποσοστό των ε, ναυτιλιακών μεταφορών στη Σκανδιναβία, εάν αμέσως ε, πλήξουμε τους ε, ιδιοκτήτες των πορθμίων, μπορεί να υπάρξει μία μετακίνηση του μεταφορικού μέτρου, άρα χρειάζεται να υπάρξει κάποια διόρθωση. Ε, ίσως όπου υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με τις οδικές μεταφορές επειδή ερχόμαστε ε, το, στην εποχή του χειμώνα καλό θα ήταν να επιβραδύνουμε λιγάκι την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων αλλά αυτό καταρχήν και θα επανέλθω μετά. Ο κύριος ε, Κέλλον. Ελπίζω να μην σηκώσετε τα φρύδια σας και στη δική μου περίπτωση. Θέλω να ευχαριστήσω ε, την κυρία Σατουχάση για όλη την προσπάθεια αυτή που κατέβαλε, η οποία είναι θετική και έχει ζητήσει να εμπλακούν όλες οι ομάδες και οι σκιώδεις εισηγητές ε, στο τελικό αποτέλεσμα. Την ευχαριστώ λοιπόν. Πριν σχολιάσω την πρόταση της Επιτροπής θα ήθελα να πω ότι ε, στηρίζω την πρώτη συμφωνία του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας και δεν θα πρέπει η, η, Επιτροπή να το διαλύσει ή να το ε, χρυσώσει. Το στηρίζουμε, αλλά όπως είπαμε πρέπει να... Ε, μεταφερθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν ξεπεράσουμε τα όρια αυτής της συμφωνίας. Όσον αφορά την ε, πρόταση της Κομισιόν, είμαι υπέρ της ευθυγράμμισης ε, των, ε, ε, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, το παράρτημα 6 της Μάρπολ για τις εκπομπές, γιατί θα βοηθήσει και την ποιότητα της ατμόσφαιρας και την ανθρώπινη υγεία. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι η απέτηση να χρησιμοποιηθούν αυτά τα καθαρότερα καύσιμα θα σημάνουν σημαντική αύξηση του και ε, όπως είπε και ο Κρίστοβε, ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην ενθαρρύνουμε ε, μια αντίστροφη μετατόπιση του μοντέλου, ένα reverse model shift όπως αναφέρεται και να επιστρέψουμε στις χερσαίες μεταφορές. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι ναυτιλιακές υπηρεσίες θα πρέπει να συνεχίσουν στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει το κατάλληλο καύσιμο. Θα ήταν παράλογο να, διακοπούν, να διακοπεί η λειτουργία αυτού του σημαντικού τομή, τομέα αν δεν υπάρχει διαθέσιμο, δηλαδή είναι κάτι εκτός ελέγχου του. Αυτό είναι κομμάτι της συμφωνίας με τον ε, Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας και πρέπει να το στηρίξουμε. Ένα άλλος παράγον που ε, ε, δεν με έχει ικανοποιήσει ακόμα είναι σε σχέση με το κόστος και το θέμα της παρακολούθησης. Δηλαδή ακόμα δεν έχω ξεκαθαρίσει πώς αναμένεται ότι θα γίνει η επιπλέον παρακολούθηση για να εξασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιείται το σωστό κάψιμο στο σωστό σημείο. Και βεβαίως η η δυνατότητα εφαρμογής, η επιβολή της εφαρμογής είναι βασικό στοιχείο. Και βεβαίως η ΣΑΤΟ ανέφερε στο θέμα στην έκθεσή της το θέμα του εάν θα πρέπει να επεκταθεί η ισχύ από τις βόρειες ακτές της Βαλτικής στις ακτές της Μεσογείου. Συνήθως προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ισότητα. Λόγω όμως των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τώρα κάποια από τα κράτη του Νότου, ίσως δεν θα, θα πρέπει να διαρωτηθούμε αν θα πρέπει να επιβάλλουμε αυτές τις ε, αρκετά δαπανηρές απαιτήσει στους, στο, ε, ε, στις περιοχές αυτές. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. uh, speaker Ο επόμενος ομιλητής Σαμπίνε Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Σάτου Χάση για την εξαιρετική έκθεσή της. Εγώ ε, προέρχομαι από το Αμβούργο που έχει ένα μεγάλο λιμάνι και λόγω της ιστορικής ε, δομής ε, του λιμανιού είναι στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή μέρα και νύχτα περνούν τα πλοία μέσω του κέντρου της πόλης και υπάρχει ρήπανση του αέρα ε, και του περιβάλλοντος ε, και ε, δεν μιλάμε όμως εδώ μόνο για τους κατοίκους των ακτών αλλά και της ανοιχτής θάλασσας ακόμη και στην Αρκτική όπου υπάρχει επιδίνωση της κατάστασης λόγω του θιαφιού που περιέχουν τα σωματίδια και γι' αυτό θεωρώ ότι η έκθεση της Σάτου Χάση είναι ικανοποιητική, οι οριακές ε, τιμές ε, είναι επίσης σημαντικές και θέλω να τονίσω ότι συμφωνώ οι οριακές τιμές να ισχύσουν από το 2015 όπως προτείνει διότι πολλές φορές μιλάμε ε, για μέτρα τα οποία θα ισχύσουν μετά από 10-15 χρόνια. Έχω μεγάλη κατανόηση για το γεγονός ότι η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να προσαρμόσουν την νομοθεσία αλλά να υπάρχουν προτάσεις όπου θα ισχύσει μία νομοθεσία από το 2020 και αργότερα είναι κατά τη γνώμη μου κάτι απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε εδώ και τρία χρόνια. Το, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει ε, αποδεχθεί Άρα βέβαια πάντοτε είναι δύσκολο να έχουμε πιο αυστηρά μέτρα διότι πιο αποδοτικά πλοία δεν μπορούν να κτίσουν όλοι και μιλάμε εδώ για να κάνουμε την Ευρώπη ε, το επίκεντρο της ε, καθαρής ναυτιλίας το θεωρούμε όμως ότι έχουμε ακόμη τρία χρόνια μέχρι ότου ε, επιτύχουμε το στόχο για την περιεκτικότητα σε θιάφη και υπάρχουν και τα φορτηγά. Θα μπορούν λοιπόν τα δηληστήρια να χρησιμοποιήσουν το ε, χρόνο που έχουν για να προσαρμόσουν τα ε, καύσιμα τα οποία προσφέρουν ε, ότι θεωρώ ότι πέραν αυτού με τις ε, τεχνικές τις οποίες προτείνουμε θα παραμένουν κατάλοιπα και πρέπει και να τις εξετάσουμε θεωρούμε ότι το καλύτερο είναι να υπάρχει μία επέμβαση στην αρχή της καύσεως για να μην μπορεί να διαφύγει το θιάφι στο διοξίδιο του άνθρακος οπότε ας μην συζητάμε μέτρα που θα εσχίσουν του Αγίου ποτέ και να επικεντρωθούμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο διότι δεν είναι σωστό οι εκπρόσωποι των ε, επιχειρήσεων πάντοτε να ε, πανέρχονται και να καθυστερούν ε, και να αναβάλουν τις εφαρμογές τις οποίες επιζητούμε διότι η καινοτομία χρειάζεται την επέμβαση του νομοθέτη για να μπορέσει να υπάρξει καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου. Ευχαριστώ. Είχαμε τον τελευταίο των σχεδόν εισηγητών και τώρα περνάμε στους υπολείπους. Δύο λεπτά μόνο. Ο κύριος Κυλακάκης είναι πρώτος. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Σάτου Χάση και να πω ότι σε αυτή την περίπτωση ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας έκανε μια αποτελεσματική πρόταση. Ε, μιλάμε για σημαντική μείωση και πρόκειται και για μια σημαντική μείωση η οποία θα γίνει και στις κατάλληλες περιοχές. Υπάρχουν βέβαια κάποιες περιπτώσεις τις οποίες θα πρέπει να ε, πιέσουμε και για πιο φιλόδοξα περιβαλλοντικά μέτρα, αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να είμαστε λίγο πιο συμμαζεμένοι και νομίζω ότι αυτή είναι μία εξ αυτών. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας αυτή τη στιγμή ασχολείται επιπλέον και με τα θέματα διοξιδίου του άρθρακα και αλλαγής του κλίματος και το μήνυμα το οποίο θα αποστείλουμε εάν προσπαθήσουμε να έχουμε ένα πολύ πιο φιλόδοξο νομοθέτημα είναι να υπάρχει λιγότερο φιλόδοξη νομοθεσία και λιγότερο φιλόδοξη πρόταση για το διοξίδιο του άνθρακα προκειμένου να μπορούν να έχουν μια καλύτερη διαπραγματευτική θέση εάν αλλάξουμε στάση εμείς σε αυτή την περίπτωση. Ε, και μάλιστα δεδομένου ότι έχουν κάνει μια πολύ λογική πρόταση και συμφωνία. Υπάρχει επιπλέον το ζήτημα του περαιτέρω κόστους. Περιοχές που έχουν πάρα πολλές ε, νήσους, παραδείγματος χάρη χώρα μου, η Ελλάδα, που έχει ε, χιλιάδες νησιά, η επιπλέον επιβάρυνση, εάν είναι πιο φιλόδεξα τα πράγματα, θα ε, τη τις ζωές των ανθρώπων. Θα περικοπούν οι μεταφορές που είναι και ζωτική σημασία για αυτούς και θα πρέπει να το υπενθυμίσουμε αυτό. Όσον αφορά τώρα το θέμα υγείας που έθιξε ο Κρίστοφερ, ευχαριστώ πολύ ε, για αυτό που είπες, αλλά πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή ο οικονομικός βραχνάς είναι πολύ σοβαρότερο πρόβλημα υγείας για τους ε, Έλληνες από τις εκπομπές ε, του διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιούζο τώρα. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την εισηγη... τη συντάκτηρα της χρωμοδότησης και τους κοιόδης εισηγητές και να ε, πω κάποια πράγματα. Η οδηγία αυτή επικαιροποιεί την οδηγία του 1999 και το, ε, τη συμμορφώνει προς το πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Θεωρώ ότι η πρόταση είναι αρκετά καλή. Η κυρία ε, Χάση ε, θέλει να πάει ε, πιο πέρα και θέλει να τροποποιήσει και το θέμα των περιοχών ελέγχου. Οι περιοχές ελέγχου είναι συγκεκριμένες περιοχές και έχουμε και προστατευμένες περιοχές και δεν πρέπει να προσπαθούμε να τα ομογενοποιήσουμε όλα σε όλες τις περιπτώσεις. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας φαίνεται λογική, διότι μας συμμορφώνει με μια διεθνή συμφωνία και νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και το εξής. Καταρχάς, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αύξηση του κόστους ε, θα πάει από το 1% στο 4% για τα δηληστήρια το κόστος του καυσίμου θα φτάσει σε αύξηση 5%. Τα διάφορα άλλα ε, κόστη θα αυξηθούν μέχρι το 40%. Αυτά όλα προκύπτουν από μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιπλέον βάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι τομείς που θα πλαχθούν περισσότερο είναι οι τομείς χαμηλής ε, ε, προστιθέμενης αξίας όπως για παράδειγμα η χαρτοβιομηχανίας, ε, και τομείς του Χάλιβα. Πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα πληχθούν και θα το ε, πληχθούν η μεταλλουργία, ε, τα, η παραγωγή χημικών προϊόντων. Και για όλους αυτούς τους λόγους θα ήθελα να πω ότι δεν συμφωνώ με την πρόταση της κυρίας Χάση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Καρτφάινς Φλόρενς. Σαν του Χάσης ευχαριστώ. Έκανες ε, μία πολύ ε, φιλόδοξη πρόταση αλλά δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή. Κάπου στην Ευρώπη πρέπει να την ε, εφαρμόσουμε εν ευθέτω χρόνο. Αλλά υπάρχουν ακόμη ορισμένα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν αλλά όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν στο σωστό πλαίσιο. Ε, να αποφύγουμε δηλαδή στρεβλώσεις ανταγωνισμού και να έχουμε ε, πιο δίκαιο ανταγωνισμό και δεν ξέρω εάν αυτή η πλήρης απελευθέρωση είναι η σωστή οδός. Τώρα, ε, το γεγονός ότι τα καύσιμα των πλοίο να είναι εκατοντάδες φορές πιο βρώμικα από ότι αυτά που χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητα αλλά ζητάτε να γίνει τώρα άμεσα η ρύθμιση και βελτίωση μόνο για ορισμένα είδη πλοίων όσον αφορά τα επιβατικά και όχι για άλλα είναι κάτι για το οποίο θα ζητούσα να μου δώσετε επεξηγήσει. Επίσης, τι γίνεται με τα, τα πλοία τα οποία φτάνουν σε μία χώρα όπου δεν υπάρχει το συγκεκριμένο καύσιμο. Το ίδιο συμβαίνει με την αμόλυβδη βενζίνη. Το είχαμε αντιμετωπίσει. Υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό τον προβληματισμό. Ευχαριστώ. Τελικά. Κύριε Σταταρέλα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να συγχαρώ και εγώ την συντάκτρια της χρωμοδότησης για τη δουλειά της. Αλλά παρά το γεγονός ότι θεωρώ απόλυτα αποδεκτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επί της ουσίας ε, συμμορφώνει την Ευρωπαϊκή Επικράτεια με μια διεθνή συμφωνία, είμαι μάλλον επιφυλακτικός ε, από τις με τις προτάσεις της κυρίας ε, Χάση. Στην Επιτροπή εδώ όλοι ανέκαθεν εκτιμούσαμε την δέσμευση και την κοινή η λογική της ε, συντάκτρας της γνωμοδότησης. Θα ήθελα λοιπόν να σας επιστήσω την προσοχή και εσάς και τους ουσκιώδεις εισηγητές να ξαναδείτε λίγο τις τροπολογίες που επεσήμανε η συντάκτρια. Τη 12, τη 14 και την 15. Οι επιπτώσεις αυτών των τροπολογιών για τον ε, τομέα ε, της ε, ναυτιλίας θα είναι πολύ ρε. Επίσης, το να περιορίσουμε το διάστημα σε πέντε χρόνια, είναι προφανές ότι τα πέντε χρόνια είναι καλύτερα από δέκα χρόνια, αν γινόταν η αλλαγή και του χρόνου ακόμα καλύτερα. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ε, ζημίες που θα προκαλέσουμε σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει λοιπόν στο σημείο αυτό και για την επέκταση στα χωρικά ύδατα θα ήθελα να ζητήσω ε, εν είδη συμβιβασμό από τους χειώδεις ηγετές να προσπαθήσουν να βρουν μία λύση που να είναι όσο το δυνατόν πιο ε, κοντά στην πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την πολύ σημαντική αυτή προσπάθεια που κατέβαλε. Αυτό είναι κάτι που απαιτεί υψηλού στόχους και στην αρχική πρόταση θεωρώ ότι υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα τα οποία ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Πρώτον, το γεγονός ότι αυτό αφορά μόνο κάποιες περιορισμένες περιοχές στη Βόρειο Θάλασσα και τη Βαλτική. Ε, είμαι πολύ υπέρ της πρότασης της εισηγήτριας που διευρύνει την ε, περιοχή στο σύνολο της Ευρώπης. Επίσης υπάρχουν προβλήματα, Ευρώπης, ε, προβλήματα υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει ως Ευρώπη να προσπαθήσουμε να είμαστε εξίσου ανταγωνιστικοί ε, σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης και όχι μόνο στη Βόρειο Ευρώπη. Αυτό θα επηρεάσει κάποιους κλάδους και κάποιες βιομηχανικές δραστηριότητες. Το άλλο θέμα που με απασχολεί είναι το θέμα της μεταβατικής περίοδου. Πρέπει κανείς να ε, μιλάει για το ιδανικό, ότι όλα μπορούν να γίνουν πολύ ε, γρήγορα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Χρειαζόμαστε αυτό το διάστημα για την οικονομία, αλλά και για να φροντίσουμε ότι το επίπεδο των εκπομπών πρέπει να επιτευχθεί. Δεν είναι ρεαλιστικό να λέμε ότι μέχρι το 2015 παντού θα υπάρχει κατάλληλη τεχνολογία. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε αυτό το θέμα, όπως επίσης και να δώσουμε και την ευελιξία, ώστε να μπορέσουν όλοι να παρέμβουν. Η δάλωση εναλλακτική θα είναι ότι θα πρέπει από τις ε, θαλάσσιες μεταφορές να περάσουμε στις χερσές, πράγμα που δεν θα είναι πάντοτε καλά. Ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι πρέπει να καθαρίσουμε τα κάσιμα των πλοίων. Ε, είναι σήμερα 2.700 φορές πιο βρώμικα από τα καύσιμα των οδικών μεταφορών. Ακόμη και αν τα νέα συμφωνηθέντα όρια τεθούν σε ισχύ, τα καύσιμα των πλοίων θα εξακολουθούν να περιέχουν από 100 έως 500 φορές περισσότερο θείο από τα καύσιμα των οδικών μεταφορών. Αυτός είναι και ο λόγος που τα καύσιμα των πλοίων θα συνεχίσουν να είναι πολύ φθηνότερα από τα καύσιμα των οδικών μεταφορών. Έτσι, το επιχείρημα ότι πολλή, ε, πολλή κίνηση θα μετακινηθεί από τη θάλασσα στη στεριά, αν τα καύσιμα των πλοίων γίνουν πιο ακριβά ως αποτέλεσμα των νέων κανόνων, είναι μάλλον μια κενή απειλή. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, η ναυτιλία να μπορεί να ανταγωνιστεί μόνο με βάση ένα βρώμικο καύσιμο. Οι περισσότερες εκπομπές των πλοίων προκαλούνται κοντά, αρκετά κοντά σε στεριά και η ρήπανση προκαλεί σοβαρές βλάβες στη δημόσια υγεία. Η μελέτη ε, από το Κέντρο Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δανίας είναι πρόσφατη αυτή που διαπίστωσε ότι οι εκπομπές ρήπων των πλοίων προκαλούν περίπου 50.000 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη. Σίγουρα υπάρχει κόστος καθαρισμού και η ναυτιλία για χώρες σε κρίση όπως η Ελλάδα είναι σημαντικό μέγεθος. Όμως ε, για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και για τις άλλες βιομηχανίες που ρηπαίνουν ήδη απαιτείται ο καθαρισμός των καυσαερίων τους. Η μείωση των εκπομπών από τα πλοία είναι πραγματικά ένας από τους φθηνότερους τρόπους για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Άλλωστε, για τα αυστηρότερα πρότυπα που πρόκειται να εισαχθούν το 2015, τα ωφέλη για την υγεία και μόνο είναι 27 φορές περισσότερα από το κόστος της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Είναι σαφές ότι πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα από τη Διεθνή Συμφωνία του IMO. Ευχαριστούμε. Ε, next speaker is from the Transport Committee, I think. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Κούν από την Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Χάση για την έκθεσή της ε, και θα πρέπει όσον αφορά την πρακτική πλευρά των καυσίμων που περιλαμβάνουν θιαφή να το εξετάσουμε διότι ε, θα πρέπει να ε, μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ναυτιλία ε, μικρών αποφάσεων, αποστάσεων να υπάρχει μία δίκαια κατανομή των βαρών και αυτό όταν το κοιτάμε στη Βόρειο Ευρώπη που έχουμε τη Βόρειο Θάλασσα, την, ε, τα κανάλια, βλέπουμε πόσο, ε, πόσες διελεύσεις έχουμε ε, εις τα πορθμία τα οποία χρησιμοποιούν δίζελ σαν καύσιμο και πρέπει να αναρωτηθούμε τι στρεβλώσεις ανα ανταγωνισμού θα δημιουργηθούν. Πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη και τον οικονομικό παράγοντα, να μην δημιουργηθεί δηλαδή το αντίθετο, δηλαδή από την αυτιλία μικρών αποστάσεων και από τη θάλασσα οι μεταφορές να μετακινηθούν στην ξηρά που θα είχε πολύ περισσότερες ζημίες και για την υγεία των ανθρώπων και οικονομικές και για την ναυτιλία και για τον ανταγωνισμό. Πρέπει λοιπόν ε, το 3,5% του θιαφιού που περιλαμβάνεται στα ναυτιλιακά καύσιμα να εξεταστεί. Για να δούμε, αυτό μπορούμε να το μειώσουμε στο 1%. Μπορούμε να το πετύχουμε και να πάει και στο 0,5%. Παρακάτω όμως τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα και παρακολουθώντας τα φρύδια του Προέδρου τον παρακαλώ να μην κάνουμε λάθη και να αποκαταστήσουμε τις ίσες συνθήκες ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Ο κύριος Περέλο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκθεση της ε, συναδέλφου του Χάση και την ευχαριστώ για τη δουλειά της. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά αυτά που είπε και ο συνάδελφος Ταταρέλα, τις τροπολογίες 12 και 14 κατά σύμπτωση εκεί όπου διαγράφεται το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναφέρεται δηλαδή στα σκάφη ε, τα οποία είναι στις ε, συνήθεις ε, γραμμές. Το θέμα είναι ότι τα πορθμία και η αναφορά ε, σε αυτά τα συγκεκριμένα σκάφη ε, διευρύνει την υπηρεσία και υποχρεώνει τα κρουαζιερόπλαια να χρησιμοποιούν ένα πιο ε, επιζήμιο καύσιμο και δημιουργούν προβλήματα και δεν τηρούμε τα όσα προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας. Αυτό το 0,10% επίσης στα καύσιμα δικαίως χρησιμοποιείται για να μειώσουμε τις εκπομπές ε, των ferry boat, τα οποία είναι πιο ρηπογόνα. Και περιλαμβάνουμε και τα σκάφη που φτάνουν στους λιμένες και συμπεριλαμβάνονται και τα κρουαζιερόπλια. Ενώ η τροπολογία της ε, εισηγήτριας θα υποχρέωνε και τα σκάφη που δεν χρησιμοποιούν ε, που δεν συγγνώμη, λειτουργούν στι συνήθει γραμμέ και στα κρουαζιορόπια που θα χρησιμοποιούν έτσι πιο πανηρό καύσιμα για όλη του τη διαδρομή. Και η αλλαγή αυτή θα δημιουργήσει μόνο αύξηση τους κόστους ε, για τα κρουαζιερόπλια και φυσικά θα είναι και πολύ σημαντικό και για τους καταναλωτές στη συνέχεια. Καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος της οδηγίας είναι να ε, έχουμε ιδιαίτερη μέρημνα για τις περιοχές ελέγχου των εκπομπών του θείου, αλλά τα κρουαζιερόπλια πολύ συχνά κάνουν πολύ μακρά ταξίδια ε, και διπυρωτικά πριν φτάσουν στους λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως ούτως ή άλλως ε, πρέπει να ε, τηρούν ε, τον κανόνα του 0,10% στο στην περιοχή ελέγχου. Να δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας παρακαλώ όσο καθυστερήσετε θα καθυστερήσει και η παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο θέμα. Θα είμαι πολύ σύντομο από, και από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Χάση για το έργο της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μελετήσουμε την ε, ανάλυση της έκθεσης. Η κυρία Χάση επανειλημμένως ε, επεσήμανε κάποια ε, χρέη ε, που υπάρχουν στα πλοία και υπάρχουν και από άποψη, ε, από άποψη ατμοσφαιρικής μόλυνσης. Πρέπει επίσης να μην ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα έχουμε 20 κράτη-μέλη που ασχολούνται με το θέμα και όπως ξέρετε ότι το θείο είναι πρόδρομη ουσία για ε, που δημιουργεί προβλά προβλήματα. Άρα και η κυρία Χάση αλλά και πολλοί από τους προηγούμενους ομιλητές ε, συμφωνούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υποκομίσουμε πολλά ωφέλη. Συμφωνούμε ότι έγινε πολύ ε, σωστή κίνηση το 2008 και είναι πολύ μετρημένη η πρόταση για να επικεντρωθούμε στην έγκαιρη εφαρμογή ε, του συμφωνίας με τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας αλλά βεβαίως και το κόστος πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όχι όσον αφορά τώρα συγκεκριμένα συγκεκριμένες προτάσεις να ξεπεραστεί το, ε, το ΣΕΚΑΣ. Δεν είχε εντολή γι' αυτό η Κομισιόν, γιατί δεν είμαστε μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Ξέρουμε ότι η κυρία Άση έχει προτείνει μία ε, δυνατότητα της, ε, του να δουλέψουμε μόνο στα χωρικά ύδατα. Πρέπει να το μελετήσουμε αυτό. Πρέπει όμως να προωθήσουμε και τις ε, ε, διατάξεις ε, του ΠΕΘ για τις ενδιάμεσες, να βρεθούν και ενδιάμεσες λύσεις. Όπως ίσως θα διαβάσατε από την έκθεση, με βάση τις διαθέσιμες μελέτες, η Κομισιόν πιστεύει ότι πράγματι υπάρχει όφελος κοστολογικό, αλλά θεωρούμε ότι δεν είχαμε την εντολή να διευρύνουμε το πεδίο και γι' αυτό πρέπει να εκφράσουν αυτή τη θέση τα κράτη-μέλη στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας στην περίοδο του 2013 που θα γίνει η αναθεώρηση. Τώρα, κάποιες ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στην ε, Επιτροπή. Ε, η εργαλειοθήκη υπάρχει ήδη από το Σεπτέμβριο. Η Κομισιόν ε, παρουσίασε το όραμά της και θέλει να συνεργαστεί περισσότερο με τα κράτη-μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διευκόλυνση της υποστήριξης της ναυτιλίας, ώστε να είναι πραγματικά βιώσιμη. Βεβαίως, μία επιφύλαξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι θα στηριχθεί το ορόσημο του 2015 συγκεκριμένα. Η προοπτική είναι πολύ πιο μακρόπνοη και αναφέρθηκαν και ε, οι στόχοι του διοξίδιου του άνθρακα. Όλα αυτά έχουν ε, σημασία. Επίσης, πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια επιστροφή στο προηγούμενο μοντέλο. Μας απασχολεί αυτό. Ε, θα παρακολουθήσουμε και πάλι την κατάσταση ε, με τους συναδέλφους της Επιτροπής Μεταφορών. Δεν ισχύει ότι μπορεί κανείς ε, να περιορίσει τις οδικές μεταφορές γιατί υπάρχει η ναυτιλία των κοντινών αποστάσεων και η ποντοπόρος ναυτιλία θεωρείται ως τρόπος μεταφοράς στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Όσον αφορά την πρόβλεψη υπεραιτέρω περαιτέρω διατάξεων για, την, για να γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα και οι διατάξεις. Κάποιος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις στην αρκτικό κύκλο. Δεν έχουμε μπει σε αυτό, αλλά βεβαίως υπάρχει θέμα εκεί. Ε, με τον άνθρακα θα μελετηθεί. Ε, ε, ρωτήθηκαμε για τον ανταγωνισμό. Καλύπτονται τα οχηματαγωγά και αν έχουν πάνω από 12 επιβάτε στην τακτική τους γραμμή ε, καλύπτονται και κατά την άποψή μας αυτό καλύπτει τα περισσότερα πλοία ε, πλέον. Τώρα, η διαθεσιμότητα των καυσίμων επίση αναφέρθηκε. Δεν θεωρεί η Κομισιόν ότι η διαθεσιμότητα του καυσίμου θα, υπάρξει, θα είναι προβληματική. Παρά τα αυτά, αυτή ήταν η σκέψη μας ε, ε, για, στο ότι δεν ευθυγραμμίσαμε τα, επιβατηγά τα επιβατικά με τα πλοία ΣΕΚΑΣ το 2015 άμεσα για να αποφευθεί κάποιος εκνευρισμός. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, η συγγήτρια θέλει... Ναι. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους και τα σχόλιά τους. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με, την άποψη της, με βάση την άποψη της πλειοψηφίας στην Επιτροπή. Κάποια σύντομα σχόλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη διατυπώσει θέση πρέπει, ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλία. Αυτή ήταν η θέση του Κοινοβουλίου όταν συζητήθηκε η φυστάμενη οδηγία. Ελπίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση, όπως και το προηγούμενο Κοινοβούλιο και το προπροηγούμενο Κοινοβούλιο. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες των συναδέλφων του Νότου για το κόστος που θα έχει υποστεί ο κλάδος. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι ο καθαρισμός των εκπομπών από τα πλοία, ακόμα και περισσότερο από ό,τι ζητά ο Διεθνής Οργανισμός ε, Ναυτιλίας, έχει κοστολογικό όφελος και για τις χώρες του Νότου, γιατί ακριβώς προκαλεί τόσο μεγάλο όφελος στην υγεία. Όσον αφορά το κόστος της νέας τεχνολογίας και των πλυντρίδων, ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι το κόστος μειώνεται πάντοτε όταν κάτι καθίσταται υποχρεωτικό. Και όσον αφορά τα τοξικά απόβλητα των πλυντρίδων, τα οποία ανέφερε η κυρία Βίλς, μία από τις προτάσεις μου είναι η υποχρέωση προς τα λιμάνια να απομακρύνουν αυτή την ύλη και να μην την απορρίπτουν στη θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ πάντως για όλα τα σχόλια λάβω υπόψη, θα πάρω τις ε, τροπολογίες των συναδέλφων και μετά θα συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ. Η, η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 12 το μεσημέρι στι 13 Και μετά περνάμε στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξης που αφορά την οδηγία για τον θόρυβο Scott Rocket. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι ο θόρυβος είναι ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Ο ΠΟΗ λέει ότι είναι ο δεύτερος παράγοντας άγχους. Ε, έχουμε το στόχο φιλοδοξιών μας στο πρόγραμμα των έξι περιβαλλοντικών δράσεων για τη μείωση της έκθεσης στο θόρυβο και την οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Έχετε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ αναφέρεται η πείρα μας μέχρι τούδε. Ο, η οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο βέβαια δεν είναι βέβαιο ότι ε, αύξησε την ενημέρωση. Ε, ευθυγραμμίστηκαν βέβαια τα κράτη-μέλη και εθνικές αρχές. Ε, οι πολίτες συμμετείχαν πολύ περισσότερο και είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ε, που προέρχεται από το θόρυβο σήμερα από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Επιπλέον υπάρχει το πλεονέκτημα ότι χρειάζεται μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να στοχεύσουμε στις πηγές του ρήβου, όπως για παράδειγμα τα αεροδρόμια και τις μεταφορές, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε. Είναι καλά τα πρώτα στοιχεία, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Δεν μπορούμε ακόμα να ποσοτικοποιήσουμε το ποσοστό και επίσης ε, θα πρέπει να κάνουμε και αξιολόγηση για να δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο των έξι περιβαλλοντικών δράσεων και προσπαθούμε να εναρμονίσουμε τους τρόπους χαρτογράφησης θορύβου και ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε μια πρόταση γι' αυτό εντός του 2012. Τα κράτη-μέλη μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη και εφαρμογή του πλαισίου. Μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία από την οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή μέσω ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εναρμόνιση. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό σε επίπεδο κρατών μελών μεταξύ αυτών που διαπραγματεύονται τη νομοθεσία για τι πηγέ θορύβου και αυτοί που εφαρμόζουν την οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Οι ανάγκες λοιπόν αντικατοπτρίζονται στα πρότυπα που έχουμε για τα αεροδρόμια και άλλους χώρους μεγάλης παραγωγής θορύβου. Τα στοιχεία που έχουμε λοιπόν συνοψίζουν και αυτά που σας ανέφερα και άλλους τομείς. Έχουμε πέντε βασικούς τομείς που μας επεσήμασαν οι ενδιαφερόμενοι και θέλουμε να έχουμε ε, στόχους για τιμές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τιμές στις οποίες να μπορούν να βασιστούν τα κράτη-μέλη για να λάβουν μέτρα. Επίσης, θέλουμε να προσαρμόσουμε τις απαιτήσει και να μειώσουμε τα επίπεδα να φτάσουμε στα ντεσιμπάλ που προτείνει ο ΠΟΕ για την έκθεση στο θόρυβο και επίσης θα πρέπει να ενισχυθούν τα σχέδια δράσης και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα για τη διαχείριση πηγών θορύβου, τεχνικές ε, ρυθμίσεις και οποιαδήποτε προσαρμογή του διοικητικού άχθους και του νομικού πλαισίου. Αυτή τη στιγμή ε, ακούμε τις απόψεις των θεσμικών οργάνων και των ενδιαφερομένων και ελπίζουμε ε, να μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε την οδηγία εντός ε, του έτους και στα πλαίσια των προτεραιοτήτων για τις μελλοντικές δράσεις για τα περιβαλλοντικά προγράμματα θα ε, ασχοληθούμε και με τα θέματα διαχείρισης ποιότητας και τη θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρήπενση και επίσης ε, να δούμε και μέτρα τα οποία μπορεί να βελτιώσουν το ένα και ταυτόχρονα να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε και το άλλο. Ε, έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερα ωφέλη όταν έχουμε καλύτερη εφαρμογή και έχουμε πιο φιλόδοξη προστασία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και αυτό φυσικά θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί και με τα όσα έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια, διότι μπορέσατε να μιλήσετε παρά το θόρυβο που είχαμε όταν ξεκινήσατε την ε, παρέμβασή σας. Υπάρχουν ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από όσους έχουν παραμείνει στην αίθουσα. Όχι, επομένως θα κάνω εγώ ένα σχόλιο για τις αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις. Υπάρχει και η κλιματική πτυχή. Θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί γιατί ορισμένες φορές υπάρχουν πολύ υψηλέ τεχνικές απαιτήσει γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξυλία για παράδειγμα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τεχνητά υλικά για να μπορέσουμε να έχουμε τη μείωση θορύβου και πρέπει να δούμε και τι γίνεται εντό των κτηρίων και ένα από τα βασικά σημεία που είχα ε, στην πείρα μου ως ε, πολιτικός ε, στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι εντός των πόλεων υπάρχουν προβλήματα θορύβου όταν προσπαθεί κάποιος να κατασκευάσει ένα νέο κτίριο και οι πολιτικοί ορισμένες φορές τείνουν να ε, παραβιάζουν την νομοθεσία και να κατασκευάζουν κτίρια εκεί που δεν πρέπει να κατασκευάζονται. Αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται να μπορούν να κοιμηθούν καλά και να εργάζονται χωρί θορύβου και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε την νομοθεσία καταλήλω. Σα ευχαριστώ λοιπόν που κάνετε αυτή την προσπάθεια και με αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίασή μα για σήμερα. Η επόμενη συνεδρίαση 19 και 20 Δεκεμβρίου. Καλή σα όρεξη.